So, λοιπόν, Αγαπητοί συνάδελφοι, με κάποια καθυστέρηση, σας καλωσορίζω συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα καλωσορίζουμε την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής ε, Βουλής μετά από ομόφωνη επιθυμία όλων των συντονιστών ε, ε, έχουμε αυτή την ε, κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών περιβάλλοντος καλώς ήρθατε σήμερα είναι μια, μια ημέρα στις Βρυξέλλες της Επιτροπής σας και θα ανταλλάξετε τώρα μαζί μας απόψε για τα μεγάλα θέματα της ε, περιβαλλοντικής ε, πολιτικής. Ε, πρόεδρος γνωρίζει εδώ πέρα το Προεδρείο. Είχαμε και πριν από λίγο καιρό μία συνεδρίαση. Οπότε καλωσορίζω την κυρία Μπούλινγκ Σρέντερ και όλους τους βουλευτές όλων των ομάδων. Να αναφερθώ λίγο στην ημερήσια διάταξή μας. Έχουμε ε, διερμηνία σε όλες τις γλώσσες πριν, ε, πλην ιστοτικών, λετωνικών και μαλτέζικων. Όλες οι υπόλοιπε γλώσσες έχουν διερμηνία. Σημείο 2, κάποιες ανακοινώσεις. Αύριο από τις 2 μέχρι τις 3 θα εξετάσουμε τη μελέτη περί ILUC θα παρουσιαστεί αυτή η μελέτη για την ε, ε, έμεση αλλαγή εκεί πέρα στην αίθουσα ASP1H1 και μπορώ να σας πω πως η ομάδα εργασίας υγείας στο πλαίσιο της Επιτροπής μας θα συνεδριάσει 25 Μαΐου από 12.30 μέχρι 3 η ώρα και θα έχουμε το εργαστήριο περί υγείας σε όλους τους τομείς της πολιτικής. Για να προετοιμαστούμε για τη νέα στρατηγική υγείας της Ένωσης. Θα ήθελα επίσης ε, να πω πως το ηλιακό αεροπλάνο από την Ελβετία προσγειώθηκε στις ε, Βρυξέλλες ε, και θα, πά, θα πάμε να το δούμε την ε, Τετάρτη το μεσημέρι στο αεροδρόμιο. Έχουν δηλώσει αρκετοί συναδελφοί ενδιαφέρον και να υπενθυμίσω πως την εβδομάδα του Στρασβούργου την 5η ε, 9 Ιουνίου 10 η ώρα θα συναντήσουμε για πρώτη φορά την Επιτροπή Περιβάλλοντος της ε, Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης όπου είναι ο πρώην συνάδελφος ο κύριος Παπαδημούλης ο πρόεδρος και επιθυμούν να συναντηθούν ε, μαζί μας. Και άρα περνάμε σημείο 4, ανταλλαγή απόψεων με τη Γερμανική Βουλή. Χαίρομαι για τότε ότι εκπροσωπούνται όλες οι πολιτικές ομάδες ε, του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Ξέρω πως είναι πάντα μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει κανείς ε, τρόπο, τόπο συνεδριάσεως, το γνωρίζουμε κι εμείς και έχουμε κάποια θέματα τα οποία θέλαμε να συζητήσουμε και δίνω τον λόγο στην ε, κυρία Πρόεδρο της Επιτροπής ε, στο Βερολίνο. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ακούσατε σήμερα πρόκειται περί μιας πρεμιέρας. Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συναντιέται με την Επιτροπή Περιβάλλοντος ενός Εθνικού Κοινοβουλίου και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος όλων των κομμάτων και αυτό δείχνει πόσο σημαντικά είναι τα ζητήματα του περιβάλλοντος, του κλίματος και θα ήθελα αυτή η ανταλλαγή να συνεχιστεί έντονη και με άλλα κοινοβούλια γιατί θεωρώ πως πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα μπορούν να επιληθούν από κοινού. Δηλαδή πρέπει να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα. Παραδείγματος χάρη σήμερα συζητήσαμε με κάποιους επιτρόπους ε, το τι θα μπορούσε να γίνει με ένα στόχο του 30% ε, καθώς υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες είναι κάπως επιφυλακτικές και νομίζω πως τέτοια ζητήματα πρέπει να τα συζητήσουμε μαζί γιατί εμείς ε, τα πέντε κόμματα της Γερμανικής Βουλής ε, στην ομάδα περιβάλλοντος συμφωνούμε, θεωρούμε πως αυτό το 30% χρειάζεται επιγόντως για να περάσουμε σε κάποιες συζητήσεις και θεωρώ ότι αυτές θα είναι χρήσιμες. Πόσο σημαντικά είναι αυτά τα ζητήματα, φαίνεται και ζητήματα πόρων, αλλά ακούσαμε και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οικονομία και η οικολογία εξετάζονται από κοινού και βεβαίως αυτό μας χαροποιεί και εμείς αυτό θέλουμε και νομίζω πως και ο χρόνος πιέζει. να σας το τι συμβαίνει στην ε, Γερμανία. Αυτή τη στιγμή έχουν βγει εκτός 14 από το 17 ε, πυρηνικά εργοστάσια. Δεν έχουν σβήσει τα φώτα. Ε, Παρ' όλα αυτά έχουμε ένα μορατόριο επίσης για 8 πυρηνικούς σταθμούς. 87% του πληθυσμού της χώρας είναι υπέρ του συντομότερου δυνατού κλεισίματος των πυρηνικών εργοστασίων και θα έχουμε μια σειρά συζητήσεων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, στην ε, Γερμανική Βουλή να δούμε πώς θα πάμε προς τα εκεί, πώς θα έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, το ζήτημα ενεργεια αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας αλλά και το πώς θα αντισταθμίσουμε την πυρηνική ενέργεια. Υπάρχουν κάποιες διαφορές στις απόψεις, αλλά δεν υπάρχει πλέον διχογνωμία για το εάν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Και είναι θετικό, πάρα πολλοί κοιτούν το τι κάνει η χώρα μας και λένε ε, αναρωτιούνται αν θα το καταφέρουμε ή όχι, εμείς θεωρούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Θέλουμε να είμαστε και ένα είδος ε, υποδείγματος γιατί μας λένε «Α, ναι, μα τότε εξάγεται πυρηνικό ρεύμα στις άλλες χώρες». Οπότε θεωρώ πως θέλουμε πως ε, θα μπορέσουμε να έχουμε αποκεντρωμένες ανανεώσιμες φυγές ε, ενέργειες. Υπάρχουν πολλά να πούμε, υπάρχουν και πολλά στην ημερήσια διάταξη. Στρατηγική προστασία του κλίματος, στόχος του 30% στρατηγική βιομάζας, ε, αποτελεσματική χρήση των πόρων ε, και το πώς θα κατευθυνθούν προς τα εκεί και τα κονδύλια της περιφερειακής πολιτικής. Αυτά και χαίρομαι που θα συνεδριάσουμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την εισαγωγή, συνάδελφε. Το πρώτο θεματικό πλέγμα θα πρέπει έτσι να καλύψουμε. Στρατηγική για την προστασία του κλίματος. Αύριο το πρωί στις 9 θα ψηφίσουμε ως Επιτροπή εμείς για την έκθεση για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 20% και παραπάνω μείωση των εκπομπών ρήπων. Τη συζήτηση του 2008 την παρακολούθησα 2009 και τώρα το ξαναέζησα. Μπορεί κανείς να διαπιστώσει σαφώς ότι υπάρχουν αντιστάσεις για μια αύξηση αυτού του ποσοστού σε 30%. Πολλοί πιστεύουν ότι το κλιματολογικό πακέτο θα ήταν τα πάντα, ενώ είναι μόνο η αρχή. Ένα πρώτο βήμα, μια πρώτη φάση μόνο. Εμείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο συχνά έχουμε και την επιθυμία να υπάρχουν ευρύτερες πλειοψηφίες γιατί <clears throat> δεν έχουμε σε σχέση με την κυβέρνηση αντιπολίτευση εμείς εδώ κάτι τέτοιο και έχουμε και το Συμβούλιο των Υπουργών των 27 κρατών μελών απέναντί μας και από πλευράς του Πράσινου από την Ολλανδία εισηγητού για αυτή την έκθεση υπήρξε, υπήρξαν πολλά σεμινάρια, συμπόσια που διεξήχθησαν, ανοιχτές συζητήσεις που έγιναν. Αύριο το πρωί θα έλεγα θα υπάρξουν μια δεκάδα περίπου ή δεκάδες συμβιβαστικέ τροπολογίες. Έτσι γίνεται στο κοινοβούλιο μας. Έχουμε και περισσότερων κοινοβουλευτικών ομάδων συμβαστικές τροπολογίες και έτσι θα υπάρξει κάποια συμφωνία για αυτές τις συμβαστικέ τροπολογίες επανειλημμένα έχει τοποθετηθεί υπέρ του 30% το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πριν από το Κανκούν το είχαμε σε ένα ψήφισμα και μετά από την Κοπεχάγη είχαμε ένα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου πάλι από αυτού του θέματος και αύριο θα έχουμε τοποθέτηση στα 30% από το Ευρωκοινοβούλιο σίγουρα. Όμως πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτή την τοποθέτηση για το τι θα κάνουμε μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι θα κάνουν οι εμπλεκόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με μηχανισμούς από το πρωτόκολλο του Κιώτο. Η αλήθεια ποια θα είναι ότι 25% θα έχουμε που θα απαιτήσουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 5% εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους μηχανισμούς του Κιώτο επιπλέον. Αυτά είναι τα κυριότερα ουσιαδέστερα αιτήματα Παράλληλα έχουμε και η κυρία, δεν ξέρω αν θα έχετε χρόνο, αμέσως μετά θα έχουμε την Επίτροπο για το Περιβάλλον που θα προσέλθει στη συνέχεια να παρουσιάσει το πρόγραμμά της. Παράλληλα με αυτή την ανακοίνωση θα έχουμε την συζήτηση για το τι θα γίνει μέχρι το 2050. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς ποιες είναι αυτές οι φάσεις που προβλέπονται καθοδόν στην πορεία αυτή για τη μέση του αιώνα όπου 80 έως 95% θέλουμε να υπάρξει μία μείωση. Από πλευράς ε, εισηγητού που ε, έχω, έχει στήσει και βρίσκεται για να παρέμβει, θα το κάνουμε εναλλάξε. Ένας, ένας, ένας από το Ευρωκοινοβούλιο, ένας από την δική σας Επιτροπή και έχουμε και ένα άλλο θεματικό πλέγμα για τη βιοπικιλότητα. Θα έλεγα μισή ώρα να μιλήσουμε για την προστασία του περιβάλλοντος και μετά για τη βιοπικιλότητα από τους συναδέφους ε, της ε, Επιτροπής ε, για το Περιβάλλον της Ομοσπονδικής Βουλής και μετά οι προβουλευτές με αυτή τη σειρά το όνομά μου είναι Γιώσεφ Γκέρπερ. Είμαι συντονιστή τη Τσεντεού Τσεσού, στην Επιτροπή Περιβάλλοντο στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο τη Γερμανία, στην Bundestag. Θα ήθελα του συναδέλφου μα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να του να τους προσφωνήσω, Πρόεδρε, και να αναφέρω ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας που λέει 40% μείωση των αερίων θερμοκηπίου στη Γερμανία πρέπει να ισχύσει μέχρι το 2020 χωρίς όρους και προϋποθέσεις κιόλας ανεπιφύλακτα Αναμένουμε και προσδοκούμε, είναι φυσικό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεπεράσει το όριο του 20% της μείωσης. Έχουμε αριθμητικά μεγέθη της, της ε, Eurostat ε, και πιστεύουμε ότι 9 χρόνια πριν από την επίτευξη του στόχου να πετύχουμε 3% όλα και όλα παραπάνω δεν είναι κάποιο ε, πιστικό εγχείρημα ή επίτευγμα και γι' αυτό παρακαλούμε θερμά η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει ένα μήνυμα για το Durban, για τη διάσκεψη για το κλίμα. Φοβόμαστε ότι αν δεν κινητοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτύχει η διάσκεψη του Durban στη Νότια Αφρική. Όμως, να επεξηγήσω κάτι για αυτή την ομοφωνία διακομματικά στη Γερμανία. Να πω δύο λόγια. Εμείς έχουμε μια πιο αποτελεσματική και θα έλεγα φιλοπεριβαλλοντική βιομηχανία που τη βλέπουμε ως μεγάλη ευκαιρία και γι' αυτό υπάρχει μεγάλη συνένεση και συμφωνία στη Γερμανία ακόμα και όσον αφορά την πάυση της εκμετάλλευσης της ατομικής ενέργειας. Χωρίς όμως την προοπτική καλύτερης οικονομικής αποτελεσματικότητας δεν θα ήταν δυνατόν οι πολίτες μας να είναι υπέρ αυτής της αλλαγής, αυτής της μεγάλης καμπής και αυτό θα μπορούσε να ισχύει για όλη την Ευρώπη. Πιστεύουμε εμεί ότι για όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε είναι μια ευκαιρία αυτή η καμπή. Και παρακαλούμε θερμά λοιπόν να ακολουθηθεί αυτή η πορεία με κάθε συνέπεια προς το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό και 25 δευτερόλεπτα. Εξαιρετικά. Ήθελα να πω ένα, ενάμιση λεπτό, ε, το πολύ δύο, αυτά είναι τα όρια για τους αγωγητές. Chris Davis φιλελεύθερη από τους φιλελεύθερους της Μεγάλης Βρετανίας. Εγώ είμαι Chris <clears throat> είμαι συντονιστής για τους φιλελευθέρους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ξεκάθαρες δηλώσεις που έκανε η Πρόεδρό σας και εσείς για τον συνδυασμό των κομματικών προσπαθειών για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Πολλές φορές η ομοφωνία που χαρακτηρίζει την πολιτική γερμανική ζωή δεν αντικατοπτρίζεται στις συζητήσεις που γίνονται ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά ούτε και στο εσωτερικό των πολιτικών ομάδων και κυρίως στη δική μου. Εν πάση περιπτώσει η Βρετανική κυβέρνηση με απόφαση που πήρε την προηγούμενη εβδομάδα συμφώνησε με τις προτάσεις τις οποίες κάναμε Έχει έρθει ο εισηγητής για το διοξίδιο του άνθρακος και θα μας πει ακριβώς τι συμβαίνει. Θα δούμε ότι έχει υπάρξει αρκετή πρόοδος, ίσως όμως όχι τόση όσο θα θέλαμε να υπάρξει, όντας φιλόδοξη. Υπάρχουν εντάσεις στο Συμβούλιο και οι εντάσεις αυτές αντικατοπτρίζονται και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και σε επίπεδο εθνικών αντιπροσωπείων. Υπάρχει ένα ποσοστό σκεπτικιστών και σε σχέση με το θέμα της ε, υπερθέρμανσης και σε σχέση με τα επιμέρους μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις οικονομικές προοπτικές. Πάντως έχει μετακινηθεί η συζήτηση. Πολλοί λέγουν ότι ακριβώς επειδή θα πρέπει να προωθηθούν οι οικονομίες μας, θα πρέπει να επενδύσουμε στον τομέα της μείωσης του διοξιδίου και δεν μπορούμε να χάσουμε την ευκαιρία, δεν μπορούμε να περιμένουμε αδρανείς πιστεύοντας ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν μόνα τους, όχι ο κόσμος αλλάζει, η τεχνολογία μας θα πρέπει να συνοδεύει αυτές τις αλλαγές. Γάιος, Γάιος Ιούλιος Κέσαρ. Εξαιρετικό όνομα. Äh, Γάιος Ιούλιος. Και αν έχω κάποια σχέση με αυτόν τον στρατηγό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν είναι απόλυτα βεβαιωμένο. Τώρα, για το διοξίδιο του άνθρακα και τους στόχους αυτούς, όταν συζητάμε για αυτό, θα ήθελα να πω εδώ για άλλη μια φορά ότι πιστεύω είναι μια μεγάλη ευκαιρία αυτή αν δει κανείς τις τεχνολογίες και όλα αυτά συνδέονται με αυτά και ό,τι μπορούμε να πετύχουμε με αυτές τις τεχνολογίες, θα πρέπει να τα σκεφτούμε πολύ καλά όλα αυτά. Το ότι εμείς οι Γερμανοί θέλουμε να έχουμε να είμαστε το υπόδειγμα, το πρότυπο για την Ευρώπη, αλλά να μην το βλέπουμε ως μέσο πίεσης μόνο αποκλειστικά γιατί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες ευκαιρίες να πισθούν οι χώρες αυτές που είναι σήμερα πιο επιφυλακτικές και διστακτικές. Όλα αυτά συνδέονται με τις οικονομικές εξελίξεις και τις θέσεις απασχόλησης. Φυσικά συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και έχουν και σχέση και με την κοινωνική συνιστόσα στην πολιτική. Ήθελα να πω ότι θα άξιζε να προβληματιστούμε και να σκεφτούμε περισσότερα διεθνή σχέδια παγκοσμιοποιημένα σχέδια και προγράμματα να εκπονήσουμε. Είχαμε πάει με επιτροπή της δικής μας Βουλής στην Αφρική και είδαμε ότι έχουν ενωθεί αφρικανικές χώρες ώστε αυτή η πράσινη ζώνη χιλιόμετρα ολόκληρα που ε, μπορεί να ε, ενεργοποιηθεί. Παράκλησή μου θα ήταν τέτοιου είδους ε, συγκεκριμένα εξειδικευμένα σχέδια και προγράμματα που μπορούμε να πετύχουμε, να ενώνονται οι Αφρικανοί και να πετύχουμε κάτι για την προστασία του κλίματος και για την ευημερία των ανθρώπων. Φυσικά εννοώ την επισητιστική ασφάλεια αυτών των ανθρώπων. Θα πρέπει να είμαστε φυσικά πρόθυμοι ελαστικά να δράσουμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο και τέτοια προγράμματα με την αναπτυξιακή η βοήθεια και την σύνδεση με την προστασία του περιβάλλοντος να προχωρήσουμε και έτσι οι ευρωβουλευτές από κοινού να πορευτούν σε αυτή την πορεία από κοινού μαζί μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ θερμά. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουδαπέστη είχαμε την κοινοβουλευτική συνέλευση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Καραϊβικής Αφρικής και Ειρηνικού. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό στην αναπτυξιακή πολιτική και βλέπουμε στην Αφρική κάποιες χώρες το έχουν καταλάβει και θέλουν να το υλοποιήσουν. Κάποιες άλλες χώρες δεν τα έχουν κατανοήσει απόλυτα και έχουν επιφυλάξεις και είναι διστακτικές. Στη συνέχεια πήγαμε με την Επιτροπή μας στην Βασοβία για την επικείμενη, ε, επερχόμενη ε, Πολωνική Προεδρία του Συμβουλίου. Και πραγματικά από την Τετάρτη το απόγευμα μέχρι την ε, Παρασκευή η συζήτηση ήταν από του Πολωνού τα επιχειρήματα. Κοστίζουν όλα αυτά πάρα πολύ, είναι πολύ δαπανηρά, επιβαρύνουν την οικονομία μα, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Βλέπει κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών το παραλληλόγραμμο των δυνάμεων ή των αντίρροπων δυνάμεων. Οι μεν κινούνται προ τη μία κατεύθυνση, οι άλλοι προ την άλλη, αλλά είναι σημαντικό να προωθηθούν αυτά τα θέματα στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, Αναρόσμπαχ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε από τη Δανία, Άννα Ρόσμπαχ, συντονίστρια για την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών. Ναι, ναι ο πρόεδρος είπε όλα όσα ήθελα να πω, δηλαδή ότι είμαστε μεταξύ αυτών των πρωτοπόρων και από την άλλη φοβόμαστε πως δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δυστυχώς πρέπει να σας πω πως ε, η ομάδα μου αποφάσισε να ψηφίσει για ένα 25% αύριο. Για μένα είναι δύσκολο Βεβαίω Εγώ είμαι από την Δανία και θεωρούμε πως εάν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω να το κάνουμε. Αλλά να βρεθεί βεβαίω και μια ισορροπία. Ε, εντάξει, να δίνουμε το καλό παράδειγμα, να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τις βέλτιστες ε, πρακτικές, αλλά να πάρουμε και με το μέρος μας τους ανθρώπους που δεν έχουν ακόμα προχωρήσει τόσο. Και εκεί πέρα νομίζω είμαστε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μάθουμε πως πρέπει βεβαίως να δείχνουμε γενικώ πως έχουμε συνέστηση της ευθύνης με το τι κάνουμε στην Ευρώπη και να δίνουμε το καλό παράδειγμα, αλλά όπως είπαμε, ε, βλέπετε, βλέπω πως οι αμερικανικές ε, εταιρείε ε, πάνε και ψωνίζουν στην Αφρική και εγκαθίστανται εκεί πέρα ε, όπου είναι πολύ φτηνή η τιμή της εργασίας και δεν εκπληρώνεται κανένα στόχος και κάτι πρέπει να γίνει με αυτή η κατάσταση. Ναι, ναι, βεβαίως. Και βεβαίως ε, πρέπει και στην ε, Δανία κάποια στιγμή να μπορούν να παράγονται και να φτάνουν τα προϊόντα, αλλά αυτό βέβαια δεν είναι δικό σας θέμα. Ο κύριος Σφάμπε από την ε, ομάδα του S5. Ναι, είμαι ο εκπρόσωπο των Σοσιαλδημοκρατών για, προστασία, ή πολιτική προστασία του κλίματος στη Γερμανική Βουλή. Αναφέρθηκε ήδη πως ε, είμαστε διακομματικά σύμφωνοι πω θα πρέπει να έχουμε ένα στόχο 30% ε, θέλω να σας πω πως εγώ είμαι και απογοητευμένος για αυτά τα οποία διαγράφονται εδώ πέρα στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί γνωρίζουμε πως αυτό το 25% συν ε, όσο είναι δεν είναι πάρα πολύ φιλόδοξο γιατί ξέρουμε πως είχαμε το στόχο 20-20-20 εμείς θεωρούσαμε και θα θέλαμε κάτι παραπάνω από τη Γερμανία η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά πρέπει να αποφασίσει αν βλέπει αυτή την ενεργειακή αλλαγή ως ευκαιρία ή όχι. Εμείς θεωρούμε πως δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, δηλαδή το εάν θα συζητάμε τα προβλήματα σε ένα υψηλό επίπεδο, αν θέλετε, κλιματική αλλαγής ή σε ένα άλλο χαμηλό επίπεδο για την ενεργειακή επάρκεια κτλ. Και αυτό νομίζω πως είναι μια ευκαιρία όχι μόνο για τη Γερμανία που το θεωρούμε ως μια οικονομική ευκαιρία, αλλά νομίζω πως και για άλλες χώρες στον κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω θα πρέπει να οργανωθεί αυτή η διαδικασία της μετάβασης στις χώρες και το λέω και ως σοσιαλδημοκράτης πρέπει να φροντίσουμε και αυτούς που δεν μπορούν τόσο γρήγορα να ακολουθήσουν αυτό το μετασχηματισμό και να οργανωθεί εντός της Ένωσης μια πολιτική για τις χώρες εκείνες που έχουν προβλήματα ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη να λάβουν την απαραίτητη βοήθεια. Παρ' όλα αυτά θεωρώ πως είναι σημαντική μια φιλόδοξη πολιτική. Γι' αυτό είμαστε σαφώς υπέρ του 30%. Ευχαριστούμε κύριε Σφάμπε. Τώρα η σειρά του εισηγητή, του κύριου Άκχα. Τι θα ψηφίσουμε αύριο και, και γιατί. Δεν μπορώ να τα απαντήσω όλα αυτά. Ο καθένας ψηφίζει μόνος του. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα και ο καθένας τα εξέφασε από όσους μίλησαν. Ζητώ συγγνώμη καταρχά για την καθυστέρηση, αλλά είχα μια άλλη συνάντηση και δεν τα κατάφερα να έρθω Από ό,τι καταλαβαίνω όμω και από ό,τι έμαθα, στο γερμανικό Bundestag υπάρχει μια, ε, θα έλεγα, διακομματική ε, συνένεση υπέρ της Ευρώπης και υπέρ των ευρωπαϊκών μέτρων στον τομέα αυτό. Και από εκεί ξεκινάμε και εμείς σαν πράσινοι. Αν κοιτάξουμε επιστημονικά το θέμα μπορούμε να καταλήξουμε και στη δυνατότητα του 40%. Αλλά εν πάση περιπτώσει η συζήτηση γίνεται και αυτό που είχε σημασία είναι αυτά τα οποία συνέβησαν τους τελευταίους μήνες, ότι δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργαζόμαστε στα πλαίσια μιας διαδικασίας όπου η μεγάλη πλειοψηφία αναγνωρίζει ότι οι πιο φιλόδοξες κλιματολογικές πολιτικές είναι καλές για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και αυτό είναι μια μετακίνηση από τις θέσεις που ακούγαμε εδώ και λίγα χρόνια, όπου πολλοί πίστευαν ότι ή θα προωθήσουμε τα οικονομικά συμφέροντα ή την οικολογία. Το ξεπεράσαμε αυτό. Δεν ισχύει αυτή η αντίθεση πλέον. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε τα δύο, οφείλουμε να τα συνδυάσουμε τα δύο. Και αυτή η εβδομάδα είναι και η πράσινη εβδομάδα στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει μια ολόκληρη σειρά δραστηριοτήτων, πράσινων δραστηριοτήτων, για την αποτελεσματικότητα χρήση των φυσικών πόρων. Αυτό σημαίνει ότι σαν οικονομία ευρωπαϊκή οφείλουμε να προπαρασκευαστούμε σωστά, έτσι ώστε να καταστήσουμε τις πρώτες ύλε τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας αποτελεσματικές και αυτό θα είναι ωφέλιμο μακροπρόθεσμα. Το θέμα είναι αν θα πετύχουμε το 30% τελικά ή όχι να πω εδώ ότι η συζήτηση την οποία κάνουμε τη θεωρώ χρήσιμη και ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη κοινωνική συνέντευξη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να φτάσουμε σε 25% σε εσωτερικό επίπεδο. 25% μεν, αλλά είναι συνενετική η λύση, υποστηρίζεται από όλα τα πολιτικά κόμματα και υποστηρίζουμε το 25% σε εθνικό επίπεδο, σε εσωτερικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι αν πράγματι εμείς θέλουμε να δούμε τις, τα κίνητρα, τα CDM, τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν στην αγορά, τότε αυτό το 30% είναι ένα μικρό συμβολικό βήμα το οποίο μπορεί να γίνει. Και κατά κάποιο τρόπο έχει υπάρξει <clears throat> ένα κόλλημα πολιτικό στο 30% ότι δεν μπορούμε να το στηρίξουμε. Αλλά μπορούμε να υποστηρίζουμε το 25% εσωτερικά. Γι' αυτό λοιπόν ο αριθμός 30% φαίνεται ότι ξαφνικά έχει πολιτικοποιηθεί και αυτό είναι κρίμα. Αν δει κανεί ποιο είναι τα επιχειρήματα των μεν και των δε, ε, θα δει ότι όλοι υποστηρίζουμε το 25% εσωτερικά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε το τελικό βήμα για να φτάσουμε στο 30% συνολικά. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό. Υπάρχει μια συνενετική τροπολογία την οποία ονομάζουμε στην ε, ευρωπαϊκή γλώσσα μια ολοκληρωμένη ε, πρόταση τροπολογίας που υποστηρίζεται από πάρα πολλές πολιτικές ομάδες αλλά από όχι όλες και που ζητά το 30%. Οι ψηφοφορίε θα γίνουν για την τροπολογία αυτή αύριο και γι' αυτό θα ήθελα να καλέσω αυτούς οι οποίοι εσωτερικά υποστηρίζουν το 25% να κάνουν το τελικό βήμα και να πούν ότι αυτό σημαίνει 30%. Ελπίζω να υπάρξει πλειοψηφία και φυσικά σαν Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν θα χρειάζεται να δυσαρεστήσουμε το γερμανικό Bundestag και να πούμε ότι εμείς ακολουθούμε την ίδια διακομματική αντίληψη και παίζουμε τον ρόλο μας σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε περιβαλλοντικό επίπεδο τον οποίο παίζαμε και στο παρελθόν όντας πρωτοπόροι στην ομοθεσία για την οικολογία. Αυτό θα συμβεί αύριο. Είναι ένα μικρό βήμα από το 25% στο 30% συνολικά και αυτοί οι οποίοι είναι υπέρ του 25% αλλά όχι υπέρ του 30% τους εύχομαι καλή τύχη στην εξήγηση της θέσης αυτής γιατί εγώ δεν τη βρίσκω ιδιαίτερα συνεκτική. Εγώ θα φανώ συνεκτικός, θα εγκρίνω το 25% εσωτερικά και το 30% συνολικά. Αυτή θα είναι η θέση μου σαν εισηγητής αύριο. Ευχαριστούμε. Αφορά και τις μελλοντικές γενναίες και έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα μέσο για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο στόχος να σωθεί ο πλανήτης. Λοιπόν, Χερμανότ παρακαλώ στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Χερμανότ είμαι εκπρόσωπος για θέματα περιβάλλοντος και κλίματος των Πρασίνων στη Γερμανική Βουλή. Αχ για την Ευρώπη και αναστενάζοντας αν δει κανείς τι κάνει η Ευρώπη δεδομένης αυτής της κατάστασης πραγμάτων. Έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά θεσμικά όργανα που γνωρίσαμε. Μιλήσαμε με πάρα πολλούς ανθρώπους. Και αυτό που με τρόμαξε και με τρομάζει είναι αυτή η φοβία, αυτή, αυτός ο δισταγμός, η δηλία που παντού ζήσαμε και βιώσαμε. Δεν υπάρχει θάρρος και γενναιότητα εδώ. Η Ευρώπη όμω πρέπει, πρέπει να αποφασίσει ποιο ρόλο θα διαδραματίσει παγκόσμια στον 21ο αιώνα η ίδια η Ευρώπη θα περάσει στους αναπληρωματικούς παίκτες ενώ η ΙΠΑ και η Κίνα θα είναι οι κύριοι παίκτες στο γήπεδο και η Ευρώπη θα περιθωριοποιηθεί ή η Ευρώπη θέλει πραγματικά και να παίξει το παιχνίδι ως κύριος παίκτη στο μέλλον αυτού του πλανήτη, αυτού του κόσμου που θα το συνδιαμορφώνει. Για να γίνει κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο να θέσει στόχους η Ευρώπη ενώπιόν της, που πραγματικά θα είναι σωστοί και θα ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των απειλών του κλίματος του πλανήτη, τουλάχιστον 30% μείωση των εκπομπών ρήπων μέχρι το 2020. Και δεύτερον, πρέπει η Ευρώπη στη συνέχεια να περάσει στην διαδικασία υλοποίησης βήμα προς βήμα κλιμακωτά γιατί δεν υπάρχει κανένα αποτελεσματικό, αποτελεσματικό τέτοιο στόχος και τρίτον πρέπει να δράσει στην παγκόσμια σκηνή με τέτοιο τρόπο ώστε να πιστούν όλοι ότι είναι πραγματικά εμπλεκόμενος παίκτη αποφασιστικής σημασίας η Ευρώπη και για ένα μικρό βήμα, με μικρά βήματα ξεκινά κανείς όπως και προτάθηκε εξάλλου να είμαστε υπέρ του 30% δεν... Είναι δυνατό σε αυτή την κοινή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ευρωβουλής και της Γερμανικής Βουλής να αποστείλουμε μια έκκληση στην ε, συνέλευση στο Κοινοβούλιο αύριο να συμφωνήσετε για αυτό το 30% στόχο. Παρακολουθείτε η συζήτηση εδώ και νομίζω το μήνυμα περνάει και είναι σημαντικό αυτό. Ο κύριος Φλόρενς, παρακαλώ, Καρλ Χάινς Φλόρενς. Ευχαριστώ για τα μαθήματα για το τι έχουμε να κάνουμε εμείς ε, στην Ευρώπη. Ως ε, μέλος της Επιτροπής πολλά χρόνια, εντάξει με ενδιαφέρουν και τα ποσοστά, αλλά βεβαίως ε, βλέπω πως σε σχέση με αυτά τα οποία αποφασίσαμε ε, κύριε Ότ, βλέπω πως ε, δεν μας ακολουθεί τόσο πολύ ο κόσμος, εάν δείτε και το Κιώτο κτλ. Βλέπετε πως οι στόχοι είναι ε, διαφορετικοί, οπότε αυτό με ενδιαφέρει εξίσου πολύ με το ζήτημα του 20%. Με ενδιαφέρει το ζήτημα με το ποια μέσα θα φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους για το εάν θα έχουμε πραγματικά δεσμευτικούς στόχους ε, για την αποτελεσματική χρήση ενέργειας, τι κάνουμε με το CDM, τι κάνουμε με όλα αυτά τα χρηματοοικονομικά ζητήματα που κινούνται γύρω από αυτό. Αυτά με, με ενδιαφέρουν, το ποια μέσα θα υποστηρίζατε εσείς για να φτάσουμε στα χύψη, στόχους και θα ήθελα να μάθω πού είναι οι δυνατότητες ελέγχου που μας δίνει το Κιώτο. Εγώ δεν είδα πουθενά τέτοιο πράγμα και είναι δύσκολο ε, σε ένα όργανο στο οποίο χρειάζεται ομοφωνία και γίνονται πάρα πολλές διασκέψεις να υπάρχει ένα όργανο τιμωρίας. Εντάξει δεν ανάγκη να είναι τιμωρία αλλά να μπορούμε να πούμε πως υπάρχει ξέρω εγώ, ένα μπλοκ που προχωράει, ένα μπλοκ που δεν ακολουθεί κτλ. Δεύτερον, εγώ θα μπορούσα εύκολα να περάσω σε ένα υψηλότερο αριθμό εάν λαβαίναμε μια απάντηση και από τα κρατη για το θέμα της αποδάσωσης. Ολόκληρη η νότιο-αμερικανική ήπειρος ε, έχει τεράστιες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και εμείς μιλάμε για κάποια νούμερα της εκατό και εκεί πέρα είναι χιλιαπλάσια ε, τα ποσά. Και βεβαίως ε, και μετά το Κανκούν είδατε τι γίνεται. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Φλίνκερτ από τους αριστερούς. Ε, ευχαριστώ. Είμαι συντονιστής για τους αριστερούς ε, στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Έχετε δίκιο πράγματι, πρέπει να δούμε πώς θα επιτύχουμε αυτό το 30% και ακριβώς επειδή εγώ είμαι από την Ανατολική Γερμανία, ξέρω το πώς ήταν η κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη και ποια πράγματα θεωρούσαμε σίγουρα και τώρα έχουμε πάλι μια νέα ε, αλλαγή. Γιατί ξέρετε πως ε, ακούγεται πάρα πολύ συχνά πως ε, ο αέρας ε, μας δίνει περισσότερη δύναμη, ε, περισσότερη ενέργεια από αυτή την οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Και ξέρετε πως ε, ειδικά σε αυτά τα σε αυτές τις ανατολικές χώρε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης θα έπρεπε να υπάρχει η κρατική βοήθεια για την ε, παραγωγή ενέργειας και για τις ε, σχετικές ε, βιομηχανίες και έτσι θα υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη αποδοχή και με μεσομακροπρόθεσμα βεβαίως ακριβώς θα αλλάξει πορεία η Πολωνία, να απομακρυνθεί από τον άνθρακα, ειδικά η Πολωνία που έχει πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό στην βιομάζα και έχει πάρα πολύ μεγάλο μέλλον εκεί πέρα και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, να μην ε, είμαστε μόνο στον τομέα των επιχειρημάτων αλλά και στον τομέα των ε, παραδειγμάτων. Νομίζω πως έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ως εθνικό κοινοβούλιο, εμείς μπορούμε να κάνουμε μόνο τα του οίκου μας και βεβαίω ε, έτσι τελείως παρενθετικά ως προς αυτό μπορούμε να δούμε και τις οικονομικές ανισότητες στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε. Με ηλιδία λίθος θα είναι ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός και τι θα γίνει με τα διαθωτικά ταμεία για την επόμενη επταετή περίοδο. Και πιστεύω πραγματικά ότι μια μετάθεση δισεκατομμυρίων πρέπει να επιτευχθεί για την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μέσα στο πλαίσιο της διαθροτικής πολιτικής για την επίτευξη των στόχων. Θα είναι πραγματικά μεγάλος αγώνας που θα δοθεί γιατί υπάρχουν και άλλες επιθυμίες από άλλες χώρες, αεροδρόμια και τα λοιπά, λιμάνια, οδικά δίκτυα, με πάρα πολύ, ας τα πω έτσι, με μεγάλη χρήση τσιμένου. Λίντα Μακέβαν παρακαλώ. Ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ όλους εδώ. Είμαι η Λίντα Μακάβαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Εργατικό Κόμμα και είμαι συντονίστρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην Επιτροπή αυτή. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ακούει κανείς το τι συμβαίνει στο ε, Γερμανικό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με τις επαφές που έχετε με κοινοβούλια άλλων χωρών γιατί όπως έχει ακουστεί δεν είναι πάρα πολύ εύκολο στο κοινοβούλιο μας να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για τις κλιματολογικές αλλαγές. Από τότε που καταλήξαμε στο νομοθετικό πακέτο το Δεκέμβριο του 2008, βλέπουμε ότι υπάρχουν συνεχείς απόπειρες για να επανέλθουμε στο θέμα αυτό σχετικά με την προτεραιότητα των κλιματολογικών αλλαγών σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα. Είναι χαρακτηριστικό το ότι είστε ενωμένοι στο κοινοβούλιο σας, αλλά εδώ στις Βρυξέλλες ένα από τα ισχυρότερα λόμπι εναντίον της καταπολέμησης των κλιματολογικών αλλαγών προέρχεται από τη γερμανική βιομηχανία που θέλει να μας πει ότι εμείς ό,τι κάνουμε βλάπτουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Γιατί υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο θέμα με τη γερμανική βιομηχανία και γιατί το μήνυμά σας δεν περνάει προς αυτούς και γιατί εξακολουθούν να υπονομεύουν τις προσπάθειές μας να νομοθετούμε εμείς εδώ. Δύο γυναίκες τέλος, Ντάγμαρ Ροτμπέρεν, τη δική μας και μετά βεβαίως έχουμε και το... την Εύα Μπουλίνγκ, ξέρετε την κυρία Πρόεδρο και μετά δεν ζήτησε κάποιος άλλο τον λόγο. Α, εσείς, Ιωζεφ. Ωραία. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Χρόνο έχουμε. Άρα Βλέπει, Ντάγμαρ, δεν, δεν θα είσαι τελευταία. Ε, δεν, δεν περίμενα να είναι τόσο απλό ούτω ή άλλω. Προσπαθώ να έχω τον τελευταίο λόγο, αλλά δεν τα καταφέρνω. Άκουσα του ε, συναδέλφους. Εγώ έλεγα πω δεν θα χρειαστεί να πω τίποτα, αλλά άμα έρχεται κάποιο και παραπονιέται, αχ, Ευρώπη, ε, εντάξει. Είμαι στην πέμπτη μου θητεία εδώ πέρα, ήμουν 15 χρόνια συντονίστρια για ολόκληρη την ε, ομάδα και θυμάμαι, η Αλόκριτη είναι επιτροπή, με συγχωρείτε, και θυμάμαι, μας λέει ο κύριος ε, Ότε εδώ πέρα να είμαστε ε, θαραλέοι. Εγώ θυμάμαι ποιοι ήταν οι θαραλέοι εδώ μέσα. Δεν υπάρχει γερμανική ε, νομοθεσία για το περιβάλλον την οποία... Περιμένετε, περιμένετε από την οποία δεν έχουμε πάει πολύ, πολύ παραπέρα. και τον κύριο Καλχαντσιλόνης. Αλλά αυτό είναι, αφορά έτσι περισσότερο το, το κλίμα και την εντύπωση που δίνεται. Ένα, ένα, ένα κομμάτι μόνο γερμανικής νομοθεσίας πήγαινε παραπέρα από την ευρωπαϊκή. Αλλιώς ε, απόβλητα, διοξίνες, ε, ε, εγκαταστάσεις καύσεων, προστασία υδάτων, ε, χωματερές, όλα αυτά είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία μάλιστα δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ εγκαίρως ε, στην Ευρώπη, κάτι το οποίο είναι πρόβλημα. Εντάξει. Τα έχω πει τόσε πολλέ φορέ σε προεκλογικού αγώνε για ευρωεκλογέ. Τέλο πάντων, να περάσουμε στην κλιματική πολιτική. Είναι εύκολο να λέμε πω είμαστε υπέρ ε, ενό 30%. Η Λίντα Μακάβαν τώρα έτσι με τον ε, βρετανικό και ευγενικό της τρόπο το είπε. Είμαστε ένα κοινοβούλιο με 27 χώρες εδώ μέσα, 27 κράτη-μέλη, τελείως διαφορετική δομή. Και έτσι με αυτές τις δομές πρέπει να καταφέρουμε κάτι το οποίο δεν θα μείνουμε ως χαρτί. Ναι, μπορούμε να αποφασίσουμε ένα 30% αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί με τις δομές που υπάρχουν σε κάθε χώρα. Και πρέπει να ομολογήσω πάντα μπαίνω στον πειρασμό να ακολουθήσω τον πιο φιλόδοξο δρόμο, αλλά τελικά αυτό το οποίο μετράει είναι να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα στην πράξη, όχι μόνο στα χαρτιά. Και δεν είμαι σίγουρη το πώς πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί η Λίνα Μακάβαν ε, που μας είπε πως αυτοί οι οποίοι ασκούν το λόμπι είναι από συγκεκριμένε χώρε για να μην περάσει το πρωτοκολλητικό, να μην εφαρμοστεί. Και πρώτα-πρώτα από τη Γερμανία και είπε και απίθυνε έκκληση να κάνετε κάτι εσείς ε, στη Γερμανική Βουλή προς τη Γερμανική κυβέρνηση. Ο ένας δίνει θάρρος και προτρέπει τον άλλο να προχωρήσει προς τα εμπρός. Έχουμε κοινό στόχο, προστασία του κλίματος. Αυτή η αμοιβαιότητα είναι καλή. Ο Ζιόζεφ παρακαλώ έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Το βρίσκω καλό να έχουμε μια τέτοια ζωντανή συζήτηση και τα επιχειρήματα να συγκρούονται και να ολοκληρώνεται η συζήτηση, διότι έτσι πραγματικά γίνεται η συζήτηση και στην κοινωνία μας και καλό είναι και εμείς έτσι να συζητάμε αυτά τα θέματα με ένταση. Συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη ότι η Ευρώπη στην κλιματική προστασία έχει επιτυχίες που μπορεί να δείξει. Για παράδειγμα, ως ηγετική τεχνολογία για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για τις ε, παρεπόμενες τεχνολογίες ε, χρήσης ε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, και σε σχέση με τη γερμανική νομοθεσία αυτή η πορεία έχει ακολουθηθεί αν μπορώ να πω και είναι νομοθεσία που είναι επιτυχής και που ξεπερνά και τα εθνικά όρια της Γερμανίας και έχει επηρεάσει και πολλά, έχει προτρέψει πολλές χώρες να κινητοποιηθούν. Αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Έχουμε προκλήσεις από άλλες χώρες σε αυτές τις τεχνολογίες, πολύ μεγάλες προκλήσεις. Κίνα που αναφέρω για παράδειγμα και για όχι υποχρεωτικά και ε, τις ίδιες κατευθύνσεις για την προστασία του, του περιβάλλοντος ε, και όσον αφορά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πραγματικά αντίπαλοι της Ευρώπης και προσπαθούν ε, να κερδίσουν έδαφος. Βλέπετε ότι μπορεί κανείς ε, να μπορέσει να ανεξαρτοποιηθεί από τα περιορισμένα καύσιμα, ορυκτά καύσιμα και οικολογικά να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας. Πρέπει με σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση και να είμαστε προπομπή, πρωτοπόροι ως Ευρώπη. Και όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο μας ως Ευρώπη, αλλά και στους άλλους στόχους για την προστασία του κλίματος. 20% που πρέπει να είναι δεσμευτικός στόχος επιτέλους για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διότι έχουμε τη δυνατότητα πιο γοργά να αναπτύξουμε αυτό το δυναμικό και να μην κολλήσουμε θέτοντας τη βιομηχανία υποπίεση. Αλλά και η κυρία Μακάβαν αυτά που είπε, έχουμε και εθνικές βιομηχανίες όπως για παράδειγμα στη Γερμανία που έχουν μεγάλες αγορές και πολλά πλεονεκτήματα μπορούν να δημιουργήσουν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 375.000 απασχόλησης έχουμε εκεί. Πριν από μερικά χρόνια ήταν 10 τόσες χιλιάδες αυτές οι θέσεις απασχόλησης. Βλέπουμε ότι δεν είναι λοιπόν αντίφαση οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η προστασία του κλίματος. Πρέπει όμως να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε ο ηγετικός ρόλος που έχουμε στην τεχνολογία στην Ευρώπη να ενισχυθεί και να μπορούμε να εξαγάγουμε. Χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες που πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ. Θα σας ευχαριστώ πραγματικά. Δεν έχει κανένα νόημα να ανταγωνίζεται κανεί να λέει ποιο έκανε καλύτερα τι και να θέλει ο ένα να θρέψει δάφνε έναντι του άλλου. Πολλέ χώρε ε, λοιπόν έχουν συνεισφέρει σε σχέση με τι τεχνολογίε αυτέ. Ο Ματία Ρόντε παρακαλώ. Ναι, η προσπάθεια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν έντονη η συζήτηση και μεγάλη η πρωτοβουλία που ξεκίνησε που από το Κοινοβούλιο Νομίζω το 1992 ήταν για το νόμο για τα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επικαιροποιήθηκε, έγινε επιτυχία, επιτυχία και σε εξαγωγές. Ξέρω γιατί πράγμα μιλώ, γιατί προέρχομαι από μια περιφέρεια που σήμερα έχουμε ένα πολύ ψηλό ποσοστό από την αιωλική ενέργεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ολική ενέργεια. Λίντα Μακάβεν ανέφερε ένα πράγμα. Είναι πραγματικά επίτευγμα το 2008 όταν είχαμε το πακέτο αυτό για το κλίμα και την ενέργεια που είχε ξεκινήσει. Λίντα Μακάβεν ήταν υπεύθυνη για το σύστημα εμπορίας τρύπων. Και μπορώ να συμφωνήσω μόνο μαζί της. Εκείνη που εκείνη που είχαν δημιουργήσει τις περισσότερες ας το πω έτσι ενέργειες εναντίον ήταν οι εκπρόσωποι των ε, γερμανικών βιομηχανιών. Παρ' όλα αυτά έγινε ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός με το πακέτο για το κλίμα και καθορίστηκαν στόχοι και αριθμητικά μεγέθη. Αν συνεισφέρουν και συμμετάσχουν και άλλοι από τις άλλες υπήρους να καταλήξουμε στο 30% και να μπορέσουμε και στο CDM και στο implementation να προχωρήσουμε. Τα τελευταία χρόνια καταδείχθηκε ότι αυτό ήταν μια ε, αδιέξοδη πορεία. Πρέπει εμείς να καθορίσουμε στόχους για τους ρήπους. Έχουμε λοιπόν αύριο την ψηφοφορία για αυτά τα θέματα. Και βρίσκω αυτά τα οποία έχουμε διαπραγματευτεί και εμπεριέχονται εσωτερικά από το 20% να πάμε στο 30% είναι ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός. Και αν αυτό το καταφέρουμε με ομοφωνία, με συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα τέτοιο ψήφισμα, μια έκθεση πρωτοβουλία είναι αυτό, δεν έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις στην ομοθεσία. Όμως, μια τέτοια έκθεση έχει μεγάλη αξία. Αν έχουμε μια ψήφιση, ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα έχουμε πλειοψηφία για περισσότερο <clears throat> επίπεδο, μεγαλύτερο επίπεδο, όταν θα καταλήξουμε στην ψήφιση κάποιου νέου νομοθετήματος και όταν έχουμε για παράδειγμα <clears throat> οχήματα τα οποία θα εκπέμπουν πολύ χαμηλούς ρήπους <clears throat> όταν έχουμε τον κίνδυνο να απειληθούν οι πλειοψηφίες ε, διότι κάποιοι συνάδελφοι θα θυμηθούν ότι έχουν βιομηχανίες ε, στην ε, περιφέρειά τους και θα θέλουν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους και πράγματα τα οποία θα θέλανε να δεχθούν μετά δεν θα μπορούσαν ίσως να περάσουν αυτά τα οποία έχουμε διαπραγματευτεί εδώ και ένα εξάμεινο πρέπει να τα σεβαστούμε και αν καταφέρουμε να πετύχουμε μια μεγάλη πλειοψηφία για αυτούς τους στόχους, τότε θα στείλουμε ένα μήνυμα, θα σηματοδοτήσουμε κάτι ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είπαμε, 30% είναι ο στόχος, αλλά έχω μεγάλες επιφυλάξεις ε, όσον αφορά το CDM και το Joint Implementation. Φαίνεται ότι δεν είναι τα σωστά μέσα, τα σωστά εργαλεία αυτά για το μέλλον. Έχετε ξεπεράσει το χρόνο, ευχαριστώ. Η κύριε ο κύριος ε, Λίμπινγκ, Τσεντεουτσέσου. Ευχαριστώ. Κάθε φορά βεβαίως που, κάθε φορά που ακούγεται ένα επιχείρημα κατά της μετάβασης ε, στις ανανεώσιμες υγείας ενέργειας μας λένε πως δεν τα δέχεται ο κόσμος, δεν δέχεται τις ανεμογεννήτριες. Να ε, σου πω ότι γίνεται στη δική μου την περιφέρεια, την εκλογική, στην ακτή της Βόρειας Θάλασσας, σχεδόν Δανία, όπου έχει πάνω από χίλιες ανεμογεννήτριες, περισσότερες από ό,τι στη Βαβαρία και τη Βάδη Βιρτεμβέργη μαζί, οπότε οπωσδήποτε και εκεί πέρα υπάρχουν διαφορές ε, εντό της Γερμανίας. Αλλά καταφέραμε να γίνει αυτό με την αποδοχή του κόσμου. Αυτή τη στιγμή βρίσκουμε και νέες εκτάσεις εκμετάλλευσης ε, του αέρα και δηλώνουν οι κοινότητες τριπλάσιες εκτάσεις ε, από αυτό το οποίο προσφέρει και το κρατήδιο, το Σλέσφι Χόλσταν. Γιατί οι άνθρωποι βεβαίως οι ίδιοι είναι και οι διοκτήτες αυτών των εγκαταστάσεων και παραμένει κάποια αξία και κάποιος πλούτος τοπικά. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποια αντίθεση μεταξύ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ε, οικονομίας, γιατί βεβαίως αυτές ήταν από τις ασθενέστερες οικονομικά περιοχές. Οπότε έτσι καταφέραμε με το θέμα αυτό να προωθήσουμε οικονομικά και αυτές τις περιοχές με αποδοχή του κόσμου που θέλει ακόμη περισσότερες τέτοιες εγκαταστάσεις. Οπότε υπάρχουν καλά παράδειγμα που μπορούν να... καλά παραδείγματα που μπορούν να μας ενθαρρύνουν σε αυτή την πορεία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να πω κάτι. Είναι καλή βεβαίως η αντίρρηση που λέει συνάδελφος. Υπάρχουν πάρα πολλά λόμπι που, λόμπι που δραστηριοποιούνται στο ευρωπαϊκό επίπεδο για το διοξείδιο του άνθρακα, για τα αυτοκίνητα και καλό είναι να συναντιόμαστε, να συζητάμε αυτά τα πράγματα και νομίζω πως θα έπρεπε να έχουμε και να έχετε κι εσείς ακόμη περισσότερες επαφές με άλλους ε, βουλευτές για να συζητήσουμε και παραδείγματα και εμπόδια και πού μπορούμε να στηριχθούμε βεβαίω. Γιατί βεβαίω υπάρχουν φόβοι, αβεβαιότητα για τις θέσεις εργασίας και που θα μπορούσε να υπάρχει μία νέα στήριξη. Και αυτό είναι κάτι που χρειαζόμαστε, γιατί όπως είπατε χρειάζεται επιγόντως και αυτό το 30% και το 40% πρέπει να φτάσουμε εκεί και το θέμα είναι πώς θα φτάσουμε. Και θεωρώ πως πρέπει να συζητήσουμε πολύ περισσότερο και να βοηθήσουμε. Αλλιώς οι φόβοι θα επεκταθούν για απώλεια πολλών περισσότερων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Και βλέπουμε πως υπάρχουν μεγάλες διαδηλώσεις σε πολλές χώρες λόγω κοινωνικών προβλημάτων. Ο κόσμος έχει σοβαρότερα προβλήματα από την ε, κλιματική αλλαγή αυτή την ε, στιγμή. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά και να τα συμπεριλάβουμε σε μια πιο έντονη ε, συζήτηση και από το που θα μπορέσουμε να βρούμε και τα χρήματα επίσης. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν το πρώτο θεματικό πλέγμα, προστασία του περιβάλλοντος και έγινε απόλυτα κατανοητό ότι η συνένεση στη Γερμανική Βουλή είναι μια ενθάρρυνση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναζητήσει και αυτό μια τέτοια ομοφωνία, συνενετικό πλαίσιο για πιο φιλόδοξους στόχους από πλευράς του. Βρισκόμαστε καθοδόν θα έλεγα αυτά που θα ψηφίσουμε αύριο αν μπορέσουν να πετύχουν στην Ολομέλεια θα είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που συζητά το Συμβούλιο Υπουργών ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει μια αμφίροπη εξέλιξη και καθοδόν προς τον Ντέρμπαν νομίζω αυτό είναι σημαντικό για τη Σύνοδο Κορυφής. Αυτή η συζήτηση να μπορέσει να συνεχίσει να μετεξελιχθεί προς το μέλλον θετικά. Η επόμενη Προεδρία θα είναι από τους γείτονές μας τους Πολωνούς. Θα πρέπει να ομιλήσουν για όλη την Ευρώπη, εξ ονόματος της Ευρώπης και όχι μόνο εξ ονόματός τους οι Πολωνοί. Θα είναι ενδιαφέρον να δει κανείς προς τα πού θα οδηγηθεί η Ευρώπη στη διάσκεψη στη Νότια Αφρική, στον Τέρμπαν. Είμαι αισιόδοξο, γιατί όπως είπα έχουμε ήδη αποφάσεις ε, από το παρελθόν και τώρα και το καλοκαίρι θα είναι σαφές ότι αν χάσουμε αυτή τη δεκαετία τότε και τους επόμενους μελλοντικούς στόχους δεν θα τους πετύχουμε. Τώρα πρέπει να επιτευχθεί αυτή η καμπή σε σχέση με τους στόχους αυτούς για το μέλλον. Ευχαριστώ, ήταν πολύ χρήσιμα και πολύ σημαντικά αυτά τα οποία συζητήσαμε. Και ε, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε κάπως χρόνο τώρα για το δεύτερο θέμα, το θεματολογικό πλέγμα η αποτελεσματικότητα των πόρων ή η βιοπικιλότητα για παράδειγμα υπό αυτό το πρίσμα. Γνωρίζουμε ότι έχουμε μια ανακοίνωση, δεν είναι ένα μέσο εργαλείο αυτό, αλλά είναι ένα έγγραφο συζήτησης. Όχι μόνο να είμαστε αποτελεσματικοί για τη συζήτηση, αλλά και για τους πόρους και η Ομοσπονδική Βουλή έχει μια ξεχωριστή επιτροπή για αυτά τα θέματα και για τα όσα τεκταίνονται σε αυτό το πεδίο. Πρέπει εμείς την Ευρώπη συνολικά στην Ευρώπη προς αυτή την κατεύθυνση να πορευτούμε και να κινηθούμε και για την Πράσινη Εβδομάδα και τις εκδηλώσεις αυτές εδώ βιοπικιλότητα είχαμε και στη μια πολύ ε, σημαντική ε, αντιπροσωπεία είχα πάει και στην ε, Νορβηγία είναι η μόνη χώρα όπου έχει ένα νομο, για το πρωτόκολλο ABS και πριν από την Ναγκόγια για το γενετικό υλικό από, τους, ε, από τα ε, νορβηγικά όρη για την ε, βιομηχανία κοσμητικών και έτσι λοιπόν με αυτό το, με αυτό το ε, δυναμικό ακολούθησε μετά η πτυχή των τροπικών δασών και από τις άλλες υπήρους η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει σε ένα νομοθετικό πλαίσιο και σε τέτοιες ρυθμίσεις ε, γιατί όλη η στρατηγική προστασία της φύσης εντάσσεται έτσι σε αυτό το πλαίσιο. Από πλευρά σας λοιπόν, Chris Davis. Ο Chris Davis ζήτησε ως πρώτος τον λόγο. Chris, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. Ανάμεσα στα θέματα της βιοπικιλότητας και τους στόχους για αυτήν είναι οι προσδοκίες που έχουμε για την αποκατάσταση των αλλιευμάτων στα μέγιστα επίπεδα αηφορίας στα επόμενα πέντε χρόνια. Ίσως δεν το πετύχουμε στα πέντε χρόνια, αλλά αυτός είναι ο στόχος. Την 13η Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Ο στόχος θα είναι η δημιουργία μιας πιο αηφόρου αντιμετώπισης του ε, φαινομένου της αλλίας. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή δημοσιευτούν οι φιλόδοξες αυτές αλλαγές αν θα τύχουν πολιτική στήριξη. Προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου υπερψηφίσαμε κατά 2 προς 1 τις, τις επιδοτήσεις προς τους αλληλείς λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων. Το να δίνουμε επιδοτήσεις σε περιόδους έλλειψης αηφορίας νομίζω ότι είναι απαράδεκτο. η πλειοψηφία των Γερμανών συμφώνησε με αυτή τη λογική. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται με τη Γερμανική Βουλή, πώς συμβιβάζεται η θέση αυτή με τη θέση της Γερμανικής Βουλής. Matthias Ματίας Μίεσ, εκπρόσωπος για το περιβάλλον του S5. Θα ήθελα να φωτίσω λίγο αυτή την πτυχή και από τη σκοπιά των επιδοτήσεων αλλά και από μια σκοπιά που δεν σχετίζεται με την αλληλεία αλλά με τη γεωργία. Γιατί αυτό το οποίο πρότεινε ο αρμόδιος επίτροπος μπορεί να αποτελέσει σημαντική συνεισφορά για περισσότερη βιοποικιλότητα, περισσότερη προστασία της φύσης. Και αυτό με το να ε, συνδεθούν οι πληρωμές ε, της γεωργικής πολιτικής σε στόχους βιοπικιλότητας, προστασίας του κλίματος, προστασίας του περιβάλλοντος ε, και συμφωνούμε στο Εθνικό Κοινοβούλιο πως αυτή η προσέγγιση του κ. Γιώλος ε, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να στηρίξουμε, να μην ανοίγουμε την κάνουλα ε, γενικώ, αλλά να συνδεθούν οι πληρωμές με κάποιους περιβαλλοντικούς στόχους. Νομίζω πως αυτή είναι μια προσέγγιση που θα μπορούσε να μεταφερθεί στην πολιτική της αλίας, ε, να συνδεθεί δηλαδή πληρώμη με κάποιους στόχους. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, πρέπει να στηρίξουμε τα επόμενα χρόνια και άρα και εμείς ως Εθνικό Κοινοβούλιο προτείνουμε να συνδεθεί η Γεωργία με τους περιβαλλοντικούς στόχους. Ευχαριστώ. Μπας Άικχαουτ. Ευχαριστώ. Για το θέμα της βιοπικιλότητας Μπορείτε να πείτε ότι δεν είμαστε στο ίδιο ακριβώς σημείο εξέλιξης με το θέμα των κλιματολογικών αλλαγών. Γνωρίζουμε τις επιπτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών, γνωρίζουμε τις λύσεις, την οικονομική αξία των λύσεων και προς τα εκεί πηγαίνουμε. Στη βιοπικιλότητα βρισκόμαστε στην φάση των γενικόλογων στόχων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποφασίσει και τι θα γίνει με την απώλεια βιοπικιλότητας το 2020. Πολύ καλός στόχος. Τι σημαίνει όμως κάτι τέτοιο. Και επανέρχομαι σε αυτό το οποίο έλεγε ο Chris Davis. Αυτά όλα σημαίνουν ότι η Ευρώπη δραστικά θα πρέπει να αλλάξει τις πολιτικές της στον τομέα της γεωργίας, της αλληλείας και αν θέλουμε να απαλλαγούμε από όλες αυτές τις βλαβερές επιδοτήσεις, τότε αυτό θα πρέπει να ισχύσει για όλες τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Θα πρέπει σαν παράδειγμα να απαλλαγούμε από το κόκκινο πετρέλαιο, που έχουμε φθηνό κόκκινο πετρέλαιο για τους γεωργούς και τους αλληλείς Γι' αυτό λοιπόν ένα επιπλέον ερώτημα προς τον Bundestag. Αν θέλουμε λοιπόν νέους νόμους για τη βιοπικιλότητα, ποια θα είναι η θέση σας όταν θα συζητήσουμε τα θέματα της ΚΑΠ ή όταν τα θέματα της κοινή αλλιευτικής πολιτικής, γιατί στους συγκεκριμένους τομείς πρέπει να υπάρξουν αλλαγές γιατί κατά τα άλλα μπορεί να συμφωνούμε σε κάποιους απόμακρους και ευγενείς στόχους, αλλά σε επίπεδο πρακτικής πολιτικής, σε επίπεδο επιδοτήσεων, αλληλείας, γεωργίας δεν αλλάζει τίποτα. Και εδώ χρειαζόμαστε τη στήριξη των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων μεταξύ των οποίων και του Bundestag έτσι ώστε τα ωραία λόγια να γίνουν σωστές πολιτικές. Γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι θα παραμείνουμε στο γράμμα και όχι στην ουσία. Γκάιος Γιούλιος Τσέζαρ της ομάδας Σεντεού θα έλεγα αν έχουμε την προστασία της βιοπικιλότητας έχουμε και εθνική στοχοθέτηση. Στην εθνική στοχοθέτηση πρέπει τα διαφορετικά συμφέροντα των ιδιοκτητών και της γεωργίας αφενός σε σχέση με την προστασία των ε, ε, ειδών της βιοποικιλότητας να συγκλίνουν οι στόχοι. Και αν συνδέσουμε τα πριμ ότι σε συγκεκριμένα μέτρα θα έχουμε συγκεκριμένες πληρωμές, θα ήταν μια καλή δυνατότητα αυτή και θα μπορούσαμε εθνικά στην δασοκομεία και στη γεωργία να συνδέσουμε τις προσπάθειες με την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος και έτσι να είμαστε πρωτοπόροι σε όσον αφορά τις όρους και οι προϋποθέσεις. Διεθνώς πρέπει να δούμε αν δει κανεί ε, το τι χάνεται από πλευράς ε, Ευρώπης, αν θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα σε σχέση με χρηματοοικονομικούς πόρους. Πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Νέα μέτρα ή ρυθμίσεις και συμβατικές υποχρεώσεις να εξετάσουμε με άλλες χώρες που σε κάποιους τομείς έχουν ήδη ξεκινήσει και προχωρούν, αλλά πρέπει να εξειδικευθούν και να εκλεπτυνθούν περισσότερο για το διοξίδιο του άνθρακα και για την προσπάθεια διατήρησης των δασών και διατήρησης της βιοπικιλότητας. Νομίζω κύριος ρόλος είναι αυτός, ένα κύριο ζήτημα όπου πρέπει μεγαλύτερες πρωτοβουλίες να αναλάβουμε. Αυτή είναι η παράκλησή μου. Ja, vielen ναι, σας ευχαριστούμε πολύ προστασία περιβάλλοντος ε, των ειδών είναι εθνικό έργο και στοχοθέτηση και όπως ε, και στην άλλη συνιστόσα πάλι και για αυτούς τους στόχους ε, που έχουμε και για αυτά τα θέματα της προστασίας ή των αλλαγών που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε μια τέτοια μικρή ήπειρο όπως την Ευρώπη υπάρχει πρόσθετη αξία αν και όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει τέτοιους στόχους και όλοι στο ίδιο πλαίσιο προσπαθούμε να υλοποιήσουμε αυτές τις υποχρεώσεις. Η Ένωση Γεωργών ήταν και εκείνη η συμμετείχε και στην Πολωνία έμαθα ότι η μισθή, η ισότητα των μισθών, αντιστοιχεία μισθών είναι ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τους Πολωνούς. Και έχουμε εδώ ένα ζήτημα, ένα θέμα όπου με τους Βρετανούς και άλλους οι, Γερμανοί έχουν, αντιμετωπίζουν προβλήματα προστασία των εδαφών. Έχουμε εδώ και το θέμα της διάβρωσης, αλλά υπό, πολλά, υπό πολλές πτυχές καλό θα ήταν να είχαμε μια οδηγία προστασίας των εδαφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι για πολλές χώρες που δεν κάνουν πολλά πράγματα ή δεν έχουν κάνει τίποτα πρέπει να δούμε ότι αξίζει τον κόπο να προχωρήσουμε, να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι. Η τροχοπέδηση από πλευράς ε, των πραγμάτων είναι δεδομένη όμως αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ. Ραλφ Λίνκορ, παρακαλώ. Ναι, η βιοπικιλότητα είναι ευρύ θέμα. Φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Τα πτηνά στα δάση στη Γερμανία έχουν ανακάμψει. Και όσον αφορά βεβαίως αυτά τα οποία χρησιμεύουν και επιτελούν κάποιο ρόλο στα λιβάδια, εκεί πέρα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Και βεβαίως η κοινή γεωργική πολιτική ε, πρέπει να φροντίσει να αποτελέσει η βιοπικιλότητα σημαντικό παράγοντα για την πληρωμή των επιδοτήσεων και να υπάρχει και μια προοπτική για τον κόσμο άρα να διαμορφώσουμε έτσι την πολιτική μας για να έχουν και ένα μέλλον οι αλληλείς για την προστασία των ε, αποθεμάτων των αλληλευτικών και να έχουν και ζωή αυτοί οι άνθρωποι γιατί αν χαθεί το ένα δεν θα υπάρχει βέβαια και καμία αποδοχή για την πολιτική. Στο σημείο αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ πως πρέπει να επέμβει πολύ ε, εντονότερα γιατί δεν θα το καταφέρουμε ως Εθνικό Κοινοβούλιο και ξέρετε πως ε, οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και λοιπές μεγάλες οδηγίες δεν θα τις είχαν περάσει σε εθνικό επίπεδο, αλλά βεβαίως πάντα ψάχνει το πιο αδύναμο κρίκο η βιομηχανία για να κάνει το λομπινγκ. Αυτό μπορεί να είναι καμία φορά το Εθνικό Κοινοβούλιο, μπορεί να είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό είναι καλή η σημερινή εκδήλωση να ανταλλάξουμε απόψεις για να μην μας παίζουν τον ένα κόντρα στον άλλον. Για να ψάχνουν βεβαίως πάντα, ξέρετε, το δρόμο της ε, ε, ελάχιστης ε, αντίστασης. Ξέρετε πως ε, υπήρχε και ένας ποταμός στη Γερμανία ο οποίος ε, πλέον ήταν βιολογικά νεκρός αλλά κάπου καταφέραμε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία τον να τον ε, αποκαταστήσουμε και ήταν κάτι το οποίο μας βοήθησε όλους. Ευχαριστώ. Η Άννα Ρόσμπαχ τελευταία από εμάς και ελπίζω σύντομη όπως πάντα. Ευχαριστώ. Και εγώ είχα πάει στην Αγγόγια βιοπικιλότητα και με θλίψη μετά συνέχεια πέρασαμε στο Μεξικό, διότι η βιοπικιλότητα με ένα πολύ μικρό εδάφιο καλύφθηκε, πολύ σύντομο. Και τελεία και παύλα, προέρχομαι από μια χώρα όπου φοβούνται τα δέντρα και κόβουν τα δέντρα επειδή ενοχλούν, λέει, ενοχλείται ο γείτονα ίσως και ξεχνάμε ότι με αυτόν τον τρόπο καταστρέφουμε και πρέπει να πω στην Ευρωβουλή Προέρχομαι από μια ευρωσκεπτιστική ομάδα, όμως στην Ευρωβουλή το θέμα των μελισσών, για παράδειγμα, το προσπαθούμε να το θέσουμε στους πολίτες και λέμε προσπαθούμε να ενωθούμε και να τα δούμε όλα αυτά από κοινού. Χρειαζόμαστε τα διάφορα φυτά ώστε οι μεγάλες ε, βλάβες που δημιουργούνται στην ε, δική μας ε, φύση να αντιμετωπιστούν και να μειωθούν. Και είναι προς το συμφέρον όλων. Αν επιτέλους ανοίξουμε τα μάτια μας και δούμε το πώς συνδέονται αυτά τα πράγματα το ένα με το άλλο συνολικά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο Φράνσιοζεφ πάλι παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Τα θέματα για τις επιδοτήσεις στον τομέα της γεωργίας και οικολογικά είναι ένα πολύ αποφασιστική σημασία θέμα όπου πρέπει πραγματικά να δούμε τις πραγματικές αναλογίες, οι ανανεώσιμες ενέργειες, που, πηγές ενέργειας που με υψηλές επιδοτήσεις μπορούν να πετύχουν. Αυτά όμως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η Διεθνής ε, ε, Επιτροπή για την Ενέργεια στο Παρίσι συνέταξε μια μελέτη και είδε και είπε ότι οι επιδοτήσεις από, ε, ε, είναι 312 δις για τα ορυκτά καύσιμα και μόνο 52 δις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα έκτο δηλαδή για τις ανανεώσιμες ενέργειες από ό,τι για τα ε, ορυκτά καύσιμα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πόσο ε, κινούμαστε για την, ε, ε, ας το πω έτσι, φθηνότερη διαθεσιμότητα των ορυκτών καυσίμων, που αυτό δεν είναι βιώσιμο, διότι δαπανούμε χρήματα των φορολογουμένων για να αντιμετωπιστούν κλιματικές αλλαγές. Και δεν είναι αυτό βιώσιμο και για την υπερχρέωση, διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν υπερχρεωμένοι προϋπολογισμοί που πιέζονται ιδιαίτερα έντονα. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ πανευρωπαϊκά αυτές οι επιδοτήσεις να τερματιστούν επιτέλους. Υπάρχουν και πολλά τέτοιες, πολλές τέτοιες επιδοτήσεις. Έχουμε και στη Γερμανία τέτοιες, την επιδότηση για τον άνθρακα ή για τους γεωργούς. Επειδή όμως αναφέρθηκε η αλληλεία, η Ισπανία για παράδειγμα δίνει άμεσες πληρωμές από τον προϋπολογισμό ώστε να είναι φθηνότερο το ως καύσιμο το ντίζελ για τους κινητήρες των πλοίων. Δεν θα πρέπει να γίνονται όμως αυτά από τις διάφορες χώρες. Πρέπει να εκπονήσουμε μια κοινή στρατηγική αυτές οι επιδοτήσεις να καταργηθούν. Αυτό ήταν και η απόφαση της λέσχης των 20, G20. Όμως ε, δεν υλοποιούνται αυτές οι αποφάσεις από πλευρά των κρατών στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Frank Schwabe. Frank Schwabe, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, αναφερθήκαμε ήδη στο πώς ε, φέρεται η Γερμανία στο ζήτημα της πολιτικής και των θαλασσών και της προστασίας ε, των εδαφών και βλέπετε εντάξει η διαφορά δεν είναι, δεν είναι ζήτημα γιατί και εδώ πέρα ο συνάδελφος κινδυνεύει να παρεξηγηθεί γιατί όταν μιλάει για Ευρώπη συμπεριλαμβάνει και εμάς ε, και εγώ Ευρωπαίος ε, αισθάνομαι, εντάξει απευθυνόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά λέω πως θα ήμουν απογοητευμένος τελικά εάν δεν φτάναμε στο 30% το οποίο είναι η ομόφωνη απόφαση στην Επιτροπή μα στη Γερμανία αλλά πράγματι υπάρχει διαφορά μεταξύ των Επιτροπών ε, και των ομάδων και βέβαια των κυβερνήσεων. Και το ίδιο ισχύει και για την πολιτική των ε, θάλασσών και της προστασίας του εδάφους και υπάρχει αντιπαράθεση με το Υπουργείο Γεωργίας. Μπορώ να πω ως Γερμανός σοσιαλδημοκράτης πως και για την πολιτική των θαλασσών και προστασία των εδαφών έχουμε και θέλουμε μια πιο οικολογική πολιτική. Γιατί βλέπετε πάμε σε πάρα πολλά ε, ζητήματα σε εθνική οικονομική πολιτική όταν μιλάμε για οριακές τιμές π.χ. στα αυτοκίνητα κτλ. Και στο Εθνικό Κοινοβούλιο συχνά έχουμε μια τέτοια κατάσταση όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε γνωρίζω πως ε, έχουν τα πράγματα και πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση για να αντιληφθούμε το πώς έχουν ε, οι πλειοψηφίες. Βεβαίως εδώ πέρα είναι τελείως διαφορετικά από το Εθνικό κοινοβούλιο, αλλά τελικά νομίζω έχουμε του ίδιου στόχους. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα δύο συναδέλφου από ένα λεπτό ο καθένα, Καλ Χάιντ Φλόρεντς. Α, εντάξει, κανονίστηκε αυτό. Όλιβε Κρίσα. Μπορώ να προσθέσω αμέσως στα σχόλιά μου στην τελευταία παρέμβαση και να πω το εξής. Στα θέματα βιοπικιλότητας η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Γερμανία πολλά οδήγησε στο να κινητοποιηθούν που εθνικά δεν μπορούσε να σκεφτεί κανείς στο παρελθόν. Natura 2000, πολλά πράγματα κινητοποιήθηκαν που εθνικά στη Γερμανία δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν. Και φυσικά συμβαίνει το ότι σε αυτό το θέμα το βιώνουμε επανειλημμένα ότι όλοι λένε ότι αυτά για παράδειγμα σε σχέση με την διάσωση των τροπικών δασών ε, όταν βλέπει κανείς στην Ευρώπη το τι κάνουμε έχουμε διαφορετική τοποθέτηση. Είναι οι άνθρωποι πιο επιφυλακτικοί. Ο κύριος Σφάμπε έχει δίκιο. Μια επίμαχη συζήτηση διεξάγεται στην ε, δική μας Βουλή. Τι πρέπει να κάνουμε, όχι τους δεκάρικους λόγους, αλλά τι συγκεκριμένα για την βιοπικιλότητα και την προστασία των ειδών πρέπει να γίνει. Συνολικά, συνολικά αυτό το θέμα της κοινή γεωργικής πολιτικής είναι σημαντικό. Όταν δει για παράδειγμα την ε, ορνηθοπανίδα κανείς, τα πιο πολλά είδη που απειλούνται είναι στις γεωργικές εκτάσεις και από μια λανθασμένη γεωργική πολιτική ο πίνακας των απειλούμενων ειδών διευρύνεται και όλα αυτά πρέπει να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε με εξειδικευμένα μέτρα. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες δράσεις σε αυτόν τον τομέα. Αυτό ελπίζω να γίνει τώρα και υπάρχουν και σκόπιμες και καλές προτάσεις ε, και προτάσεις που και πρωτοβουλίε που αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να δούμε ότι δεν είναι πάντα σωστέ οι τοποθετήσει τη γερμανικής κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω η μια μισή ώρα που συζητήσαμε ήταν πραγματικά χρήσιμο χρήσιμος χρόνος. Το, το πείραμα αυτό πέτυχε διότι έχουμε την επαφή με ένα ε, Εθνικό Κοινοβούλιο, με μια Επιτροπή Εθνικού Κοινοβουλίου, εμείς εδώ στην Ευρωβουλή, ήταν χρήσιμη η συνάντησή μας, το βλέπουμε και είναι χρήσιμο και συμφωνούμε η Ευρώπη να μπορέσει να, να ακολουθήσει την οδό προς την local economy, τοπική οικονομία για την διασφάλιση των πόρων και των προσπαθειών. Ε, όλα αυτά τα υιοθετήσαμε και τα ακολουθήσαμε και όλοι μιμούνται αυτή την πορεία βλέπουμε δισεκατομμύρια τα 7 δισεκατομμύρια σήμερα στον πλανήτη που σύντομα θα γίνουν 9 δισεκατομμύρια θα πρέπει να ακολουθήσουν μια, ένα άλλο διαφορετικό οικονομικό πρότυπο που θα βασίζεται στην αηφορία και στη βιωσιμότητα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στις Βρυξέλλες για αυτή τη συζήτηση, για αυτή τη συνάντηση. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας στο Βερολίνο όπως εσείς μας ευχόσαστε κάθε επιτυχία στο έργο μας στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστούμε και θα τα ξαναπούμε με την επόμενη ευκαιρία που θα συναντηθούμε. Αγαπητέ Τζολάιν, σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που είχαμε να είμαστε εδώ πέρα και όλους τους άλλους ε, συναδέλφους και βεβαίως ε, εμείς αποφασίσαμε ως ε, δώρο να μην σου δώσουμε έναν τόμο που δίνει συνήθως η Βουλή αλλά έναν τόμο που περιέχει κάποιες φωτογραφίες κάποιων ε, μέρων ε, τσιτόπων που θα χαθούν ε, προσεχώς λόγω της κλιματικής αλλαγής και είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι για να ξέρουμε ποιο είναι το αντικείμενό μας. Αυτό είναι λοιπόν το δώρο σου. Ευχαριστώ. Θα ρίξω μια ματιά. Είναι ωραίο αλλά θλιβερό άρα για τους ωραίους αυτούς οικότοπους και βιοστήματα που κινδυνεύουν. Έχουμε σε λίγα λεπτά την Επίτροπο του Κλίματος. Εάν έχετε χρόνο μπορείτε να καθίσετε να την ακούσετε. Αλλιώς ε, είστε επανειδήν και ε, θα τα ξαναπούμε όπως είπαμε στην επόμενη εκδήλωσή μας. Ευχαριστώ πολύ. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort. Punkt 5 der με το 5 στην ημερήσια διάταξη. Χαιρετήσω θερμά την Κόνι Χέντεγκαρντ, Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος, του κλίματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συζήτηση διεξάγεται μέσα στο πλαίσιο του διαθρωμένου διαλόγου που συμφωνήσαμε μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα εργασίας όσον αφορά τους επιτρόπους ε, για το επόμενο έτος. Βλέπω ότι οι συνάδελφοι από την Ομοσπονδιακή Γερμανική Βουλή παρέμειναν στην αίθουσα. Βλέπω ότι και ο επόμενος φιλοξενούμενος Φίλιπ Μέσταντ ε, από την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι παρόν και υπάρχει εδώ ενδιαφέρον για τη συγχρηματοδότηση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτών των προσπαθειών Κυρία Χιντεγκάρτ, σας ευχαριστούμε. Συνερχόμαστε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβούλιο για το μεγάλο θέμα προστασίας του κλίματος. Βρισκόμαστε στην ίδια πορεία και κατεύθυνση. Σας δίνω αμέσω τον λόγο. Έχουμε <clears throat> χρόνο μέχρι τις και μισή. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πάντα χαρά να είναι κανείς εδώ ανάμεσά σας Έχουμε τη δυνατότητα να συναντώμεθα συχνά, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν εξελίσσονται με ικανοποιητικό τρόπο, όπως τα θέματα τα οποία συζητιώνται αυτή τη στιγμή και σε διεθνές επίπεδο και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό και αναφέρομαι στο πρόγραμμα εργασίας. Ευχαριστώ σχετικά με αυτά που είπατε για την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011 όπως επίσης και την προετοιμασία την οποία κάνουμε για το πρόγραμμα του 2012. Κάνουμε τεράστιες προσπάθειες έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να είναι ηγέτη στην καταπολέμηση των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών και σε επίπεδο εσωτερικών και επίπεδο εξωτερικών αλλαγών, ε, πολιτικών. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να βάλει τα θεμέλια του πιο φιλόδοξου προγράμματος καταπολέμησης των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών και πέραν του 2011. Οι δύο βασικές μας, τα δύο βασικά μας επιτεύγματα είναι η υιοθέτηση του οδικού χάρτη για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών και αυτό φαίνεται και μέσα από το πρόγραμμά μας του 2011 και η συνεχής εφαρμογή του ενεργειακού και κλιματολογικού πακέτου σε σχέση με τις εκπομπές καυσερίων όπου ελήφθησαν οι αποφάσεις για τα ανώτατα όρια, τα όρια αναφοράς όπως επίσης και για τις κυβερνοεπιθέσεις. Να σχολιάσω τώρα τον οδικό χάρτη για το 2050 και το πέραν του 20% μείωση. Ξέρετε ότι υιοθετήσαμε τον Μάρτιο τον χάρτη αυτό. Το Συμβούλιο ε, Υπουργών Περιβάλλοντος στις 21 Ιουνίου προβλέπει την υιοθέτηση συγκεκριμένων ε, συστάσεων. Το πακέτο αυτό προτάσεων είναι τμήμα της ε, της ε, πρωτοβουλίας για το 2020 υποστηρίζει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 είναι οι λεγόμενες πρωτοβουλίες flagship και επίσης βλέπει και πέραν ε, του ορίζοντα του 2020 για περαιτέρω δυνατότητες μείωσης ε, κατά 80 με 95% το 2050 σε σχέση με το 2000 από το σύνολο των αναπτυγμένων χωρών. Η συνολική οικονομική ανάλυση του οδικού χάρτη δείχνει ότι για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς κατά 80 με 95% όλες οι μειώσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν σε εσωτερικό επίπεδο για να έχουμε σε εσωτερικό επίπεδο 80% στόχο. Εδώ είναι ε, θα έλεγα ένα από τα σημαντικά συστήματα αλλαγών που θα πρέπει να κάνουμε. Μακροπρόθεσμα δεν θα έχουμε πάρα πολλέ εναλλακτικέ λύσει σε σχέση με το συνδυασμό με άλλες χώρες και οικονομίες. Και αν θέλουμε να περάσουμε σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών θα ήταν σοφό από τώρα να επενδύσουμε σε τοπικό επίπεδο και όχι εμείς να επενδύουμε σε καινοτομίες σε συνεργασία με ανταγωνιστές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα χρησιμοποιήσει τον οδικό χάρτη για να ορίσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και πολιτικές πρωτοβουλίες όπως η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές, το πρόγραμμα δράσης για την ενεργειακή απόδοση που έχει παρουσιαστεί και αυτό και επίσης και ο οδικός χάρτης τον οποίο προανέφερα για το 2050. Σχετικά με την ανακοίνωση για το πέραν του 20% να πω ότι καλωσορίζω την πρόταση ψηφίσματος όπως επίσης και τις τροπολογίες. Είναι επικοδομητικές οι τροπολογίες και οδηγούν θα έλεγα σε μια κατάσταση από όλη, την οποία όλοι θα βγουν κερδισμένοι. Είναι πιθανό ε, το ψήφισμά σας να υπογραμμίζει κάποιες από τις συστάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. Αυτό πετύχαμε τους τελευταίους 12 μήνες. Όταν είχαμε προτείνει την ανακοίνωση πέρυσι το Μάιο του 20 και 30% ήταν για πρώτη φορά που υπογραμμίσαμε ότι υπάρχει εδώ ένα στοιχείο συμφέροντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοώ με αυτό. Ε, θα βελτιώσουμε την ανεξαρτησία μας στον τομέα της ενέργειας, θα βελτιώσουμε την ανεξαρτησία μας στον τομέα της της προμήθειας καυσίμων, αλλά και θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης μέσω ε, πίεσης για την ανάκαμψη της οικονομίας. Θα πρέπει να πω εδώ ότι θεωρώ θετικό ότι η μείωση του 20% ε, την κρίση σας ότι η, μείωση κατά 20% δεν είναι επαρκής και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να έχουμε υψηλότερους στόχους και να φτάσουμε στο 25% μετά το 2020 για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, αν πετύχουμε τους στόχους μας, θα έχουμε ήδη μια μείωση της εκπομπής καυσέριων κατά 25%. 5% λοιπόν επιπλέον σε εσωτερικό επίπεδο με τον στόχο του 20% τον οποίο προσπαθούμε να πετύχουμε. Ελπίζω να δεχθείτε λοιπόν αύριο την πρόταση ψηφίσματος επί τη βάση μιας ευρυτάτης πλειοψηφίας. Αυτό θα ε, ξεκαθαρίσει θα έλεγα την πορεία για την ψήφο του Συμβουλίου τον Ιούνιο και θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από πλευράς Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ETS είναι το λεγόμενο flagship ε, της, ε, η ναυαρχίδα της πρωτοβουλίας μας όλα τα μέτρα τα οποία προτείνονται. Προβλέπεται να υπάρχουν και ενδιάμεσα συνοδευτικά μέτρα. Έχουν υπάρξει κανονισμοί και για τις αποφάσεις στα επίπεδα αναφοράς. Υπάρχουν πολλά να γίνουν ακόμα για μια έγκαιρη εφαρμογή βέβαια των μέτρων αυτών. Τεχνικά εφαρμοστικά μέτρα θα πρέπει να υιοθετηθούν πριν από το τέλος του 2011 μετά από τις τελευταίες ε, προβληματικές καταστάσεις σε σχέση με τα ηλεκτρονικά μικρόα, ξέρετε ότι πήραμε ορισμένα προληπτικά μέτρα, στήσαμε επιπλέον μέτρα ασφαλείας, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά συνεχίζουμε και μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια μας. Όπως επίσης γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το επόμενο MFF για την υιοθέτηση ενός συνόλου προτάσεων μέχρι το τέλος του ε, Ιουνίου. Στα πλαίσια αυτά, το mainstreaming για τις κλιματολογικές αλλαγές είναι απαραίτητο. Αυτό αφορά κυρίως και τα ταμεία συνοχής και την πολιτική στον τομέα της γεωργίας και την έρευνα για την ανάπτυξη και τις εξωτερικές πολιτικές. Το mainstreaming λοιπόν των κλιματολογικών αλλαγών θα πρέπει να είναι απτό και ε, ορατό. Ε, πρέπει έτσι να υπογραμμίσουμε τους στόχους μετρίασης των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών και για να το πετύχουμε αυτό απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις. Επενδύσεις που θα επηρεάσουν θετικά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αυτό θα ανταποκρίνεται επίσης και στα μέτρα τα οποία θα πάρουμε στους επόμενους προϋπολογισμούς μετά το 2012. Πέραν της προετοιμασίας των τροπολογιών για τα αρχεία και τα μητρώα, ε, απαιτείται και συνεχίζεται η προσπάθεια για τον έλεγχο της αγοράς ε, των καυσαερίων του άνθρακα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν απάτες και στρεβλές συμπεριφορές στα πλαίσια της νέας και αναπτυσσόμενης αγοράς ETS. Ξετάζονται επιλογές όπως και η ταξινόμηση των επιτροπωμένων ποσοτήτων στα πλαίσια της αναθεώρησης ε, των χρηματοδοτικών μέσων και στα πλαίσια της οδηγίας επίσης για τις καταχρήσεις στον τομέα της αγοράς, για τις αερομεταφορές, η εφαρμογή της νομοθεσίας για να συμπεριληφθούν οι αερομεταφορές στα συστήματα ανταλλαγών ποσοτήτων είναι σε εξέλιξη. Όλα τα στοιχεία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο και το επόμενο σημαντικό στάδιο θα είναι η δημοσίευση στο τέλος του χρόνου των ποσοτήτων διοξιδίου του άνθρακα που θα επιτρέπεται να φτάνουν οι αερομεταφορείς. Έχουν υπάρξει τεχνικές ρυθμίσεις και τα κράτη-μέλη μας έχουν μεταφέρει ήδη υψηλά επίπεδα προσαρμογής και αυτό αφορά τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Πολιτικά όμως κάποιες, ε, κάποιοι αερομεταφορείς τρίτων χωρών εκφράζουν την αντίθεσή τους στη δράση μας. Έτσι λοιπόν, από τη μία θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη σωστή και ήπια εφαρμογή του νόμου, από την άλλη θα πρέπει να εξηγήσουμε την νομοθετική μας δραστηριότητα στις άλλες εταιρείες. Τα κοινοβούλια έχουν σε επίπεδο κοινοβουλευτικό πάρα πολλή δουλειά για να εξηγήσουν τις θέσεις μας. Περιλαμβάνονται εφαρμοστικές ε, ε, εξουσίες σχετικά με τον έλεγχο των εισερχομένων πτήσεων έτσι ώστε να λαμβάνονται αντίστοιχα μέτρα και από τις τρίτες χώρες. Δηλαδή κάτι κάνουν οι χώρες αυτές που είναι ισότιμο με αυτά τα οποία εμείς απαιτούμε και γίνεται δεκτό αυτό στα πλαίσια του υπολογισμού της πληρωμής τους. Πολλές είναι οι χώρες οι οποίες προχωρούν προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά και εδώ όταν συναντάτε ε, ε, συναδέλφους σας από άλλα κοινοβούλια να εξηγείτε λίγο την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε υπάρχουν εδώ πολύ σημαντικές αρχές που βρίσκονται σε διακύβευση και θα έλεγα ότι απαιτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει την προσπάθειά της με πάρα πολύ μεγάλη επιμονή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπογραμμίσει τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για τις κλιματολογικές επιπτώσεις των αερομεταφορών εκτός διοξιδίου του άνθρακα. Στα πλαίσια αυτά έχουμε εκφράσει την πρόθεση να αντιμετωπίσουμε τα θέματα NOx, των εκπομπών NOx. Επίσης, e και ό,τι άλλο έχει σχέση με άλλες μορφές μόλυνσης. Θα πρέπει όμως η πρόταση να βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία. Μια πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει δείξει ότι υπάρχουσα ε, επιστημονική τεκμηρίωση για τα οξύδια του αζότου, τα νόξο δεν είναι ακόμα ε, πιστική. Απαιτείται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει με μια νέα πρόταση, να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην σωστή εφαρμογή του πλαισίου για τις αερομεταφορές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων. Όπως είπα, στα πλαίσια των διεθνών διαπραγματεύσεων θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξανασυζητήσουμε όλα αυτά. Θα προσπαθήσουμε εμείς να καταστήσουμε χρήσιμο το τέρμπαν και στα πλαίσια της συνέχισης ε, της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίστηκαν στο Κανκούν. Θα περιμένουμε επίσης ε, και τις μελλοντικέ νομικές υποχρεωτικές ρυθμίσεις. Γνωρίζετε ότι τα θέματα αυτά είναι δύσκολα και περίπλοκα και γι' αυτό θα πρέπει να μην αγνοήσουμε και άλλα θέματα όπως οι ε, θαλάσσιες μεταφορές, τομιακές αντιμετωπίσεις των προβλημάτων και αερομεταφορές και άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει εμείς να θέσουμε στη διάσκεψη του Ντέρμπαν. Κάποιες άλλες πρωτοβουλίες. Θα προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής βιοκαυσίμων και βιοϊγρών θα πρέπει να υπάρξουν τεχνικές αλλαγές σε σχέση με την παραγωγή των βιοκαυσίμων επί τη βάση των τελευταίων επιστημονικών στοιχείων. Η ανταλλαγή γεών μπορεί να βοηθήσει τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων στην παραγωγή βιοκαυσίμων. Αυτή είναι μία από τα ένα από τα συμπεράσματα στο οποίο έχουν καταλήξει οι επιστήμονες. Από την άλλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει μια μελέτη επιπτώσεων και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις και στο εσωτερικό της Επιτροπής και θα τα συζητήσετε αυτά αύριο αναλυτικότερα με τις υπηρεσίες μου σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού. This is one of the σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για τα χλωριούχα αέρια, είδαμε ότι ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει δύο στοιχεία και επ' αυτής της βάσεως εφόσον χρειάζεται θα υπάρξουν προτάσεις για την τροποποίησή του. Πάντα για τα χλωριούχα αέρια. Πρόθεσή μας είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει την πρότασή της στα πλαίσια της φθινοπορεινής περίοδου και νομίζω ότι εδώ ε, απαιτούνται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προετοιμάζει μια πολύ προσεκτική έρευνα των επιλογών που έχουμε για να κάνουμε τη συγκεκριμένη πρόταση. Θα είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόταση ενίσχυσης και ισχυροποίησης του κανονισμού πριν από το καλοκαίρι του επομένου έτους. Προετοιμάζουμε την αναθεώρηση του μηχανισμού αναθεώρησης του μηχανισμού λήψης αποφάσεων για το streamlining, streamlining συγγνώμη, είναι μία από τις βασικές πρωτοβουλίες ε, του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2011 για την απλούστευση της νομοθεσίας σχετικά με τις αλλαγές χρήσης των χειών και την δασοπονία. Έχουμε συγκεκριμένους στόχους μείωσης ε, των καλλιεργειών, των εδαφών μάλλον, στα πλαίσια του συνολικού πακέτου που θα πρέπει όμως να συνοδεύεται από μια νομοθετική πρόταση και η πρόταση θα γίνει πριν το τέλος του χρόνου. Η πρόταση για το πρόγραμμα εργασίας του 2012 βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας και θα υιοθετηθεί στις 26 Οκτωβρίου. Στόχος του προγράμματος σε σχέση με τις κλιματολογικές αλλαγές πέραν των διεθνών διαπραγματεύσεων και σε σχέση με την εφαρμογή των μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια θα αντιμετωπιστεί και στα πλαίσια του οδικού χάρτη του 2050 και της περαιτέρω μείωσης των εκπομπών καυσαερίων. Τέλος, τον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας, η νομοθεσία, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά να συμπεριλάβουμε τις εκπομπές καυσαερίων του εμπορικού στόλου στους στόχους για τη μείωση των καυσαερίων αν δεν έχει πάρει ειδική διεθνή συμφωνία μέχρι το τέλος του 2011. Εμείς προφανώς και θέλουμε να υπάρξει μια διεθνή συμφωνία και θέλουμε μέτρα τα οποία να εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες. Αυτή θα είναι η καλύτερη λύση όταν μιλάμε για ένα τόσο σφαιρικό τομέα, παγκοσμιοποιημένο τομέα, την εμπορική ναυτιλία. Αλλά δεν βλέπουμε όμως τα διεθνή σώματα των Ηνωμένων Εθνών να προχωρούν σε μια κάποια συμφωνία σε σχέση με τη μείωση και ε, το να μην αναλάβουμε δράση δεν είναι επιλογή για τον τομέα της ναυτιλίας. Συνεχίζουμε λοιπόν διαβουλεύσεις με τους εμπλεκομένους σχετικά με την πρόταση που κάνουμε για τα ευρωπαϊκά μέτρα. Υπάρχει ένα, ένα πάνελ στο οποίο προεδρεύω εγώ και ο Επίτροπος Κάλλας και συμμετέχετε και εκπροσωπή δική σας. Οι υπηρεσίε μου θα κάνουν μια πρόταση κατά τη διάρκεια του 2012 που θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα φυσικά το ετήσιο για το 2012. Δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις για την εμβέλεια και τις προτινόμενε πολιτικές. Έχει ξεκινήσει διαβούλευση με τους εμπλεκομένους και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένε λύσει και προτάσει στο τέλο του έτου. Αυτό φυσικά ε, ε, είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί αφού ληφθεί υπόψη και το θέμα των επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Προσπάθειες λοιπόν για το 11 συνεχίζονται, το 12 το πρόγραμμα δεν έχει υιοθετική πλήρως, ο διαφορετικός διάλογος με το Κοινοβούλιο είναι σημαντικό χαρακτηριστικό της πολιτικής μας για τον επόμενο χρόνο. Yeah.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 Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που ήρθατε με τόσο συνολική ενημέρωση. Πρώτα απ' όλα να πω πως έχουμε καλά νέα για το iLook και αναμένουμε βεβαίως να το δούμε τον Ιούλιο το χρειαζόμαστε, αλλιώς αυτά τα οποία, αυτά τα οποία ακούγαμε πριν από λίγες εβδομάδες στο Κοινοβούλιο που διώχνουν τον κόσμο από τη γη του στην Αφρική για να καλλιεργήσουν βιοκαύσιμα, ε, θα επεκταθούν και πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στον κλάδο πως θα υπάρχουν αυστηροί κανόνες από τις Βρυξέλλες έτσι ώστε να έχουμε μόνο καλά βιοκαύσιμα που θα μετρήσουν για τους στόχους μας. Επίσης, για την ε, εκμετάλλευση πετρελαίου από την, την άμμο με πίσα. Σχιστολιστική άμμο. Ε, και για την ε, μεταρρύθμιση επίσης της σχηνή γεωρικής πολιτικής και της αλληλευτικής πολιτικής. Τι κάνετε ε, εσείς ως Γενική Διεύθυνση γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά ε, και για το κλίμα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 bei den Βρισκόμαστε και για την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Οδικού Χάρτη. ποιε αποφάσει αποφάσεις ζητείτε να λάβει το Συμβούλιο και πότε και ποιε αποφάσει θα πρέπει να εξετάσει το Συμβούλιο στο αμέσο μέλλον και ποιες επιπτώσεις θα υπάρξουν από αυτές τις αποφάσεις. Ποια θα είναι η συνέχεια που θα δοθεί. Ευχαριστούμε. Εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ήταν, Αυτό ε, ήταν μία από τις ερωτήσεις μας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ την Επίτροπο για τη σύντομη παρουσίασή της, αλλά νομίζω πως ε, γίνεται πιο κρίσιμο τώρα όχι μόνο να ξεκινήσουμε τον οδικό χάρτη για το 2050, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι πως έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε τώρα. Π.χ. το σύστημα εμπορίας εκπομπών στην αεροπορία ξεκινάει ένα λόμπι πως χρειάζεται να αλλάξει ξανά η νομοθεσία. Είναι κακό αυτό το οποίο συμβαίνει ξανά από την αρχή και συνήθως χρησιμοποιείται το επιχείρημα της οικονομικής κρίσης και νερώνουμε έτσι την ε, νομοθεσία μας και αν δείτε το οικονομικό επιχείρημα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι στην κλιματική πολιτική αλλά υπάρχει μια τάση προς την αντίστοιχη κατεύθυνση οπότε μπορείτε να είστε πιο ακριβείς πως πράγματι θα επιμείνετε στην ε, υπάρξη νομοθεσία και έχετε την υποστήριξή μας και πράγματι πως όσον αφορά τα βιοκαύσιμα πράγματι χρειάζεται ο παράγοντας iLook και όταν μιλάμε δε ε, για τα σχιστολιθικά πετρώματα που περιέχουν πετρέλαιο να μην υποκύψουμε στο καναδικό κόμπι που είναι πάρα πολύ δραστήριο και ήταν δραστήρι ε, και στην Καλιφόρνια αλλά η Καλιφόρνια δεν υπέκυψε οπότε υποθέτω πως η Ευρώπη επίσης δεν θα υποκύψει επιπλέον και βεβαίως έχουμε θέματα στα οποία θα θέλαμε φιλοδοξία, αλλά να τονίσουμε πως σας υποστηρίζουμε όταν παραδείγματο χάρη συζητάμε τα βιοκαύσιμα στην αεροπορία, πως να μετράνε μόνο εάν εκπληρώνουν το κριτήριο της αηφορίας. Και πράγματι αυτή είναι η θέση σας και σας υποστηρίζουμε. Οπότε να επιμείνετε, να είστε φιλόδοξοι. χρειαζόμαστε οικονομικά και όλα τα αντίστα επιχειρήματα που λένε περί οικονομικής κρίσης ε, δεν θα πρέπει να τα ακούμε. Ευχαριστώ. Κυρία Χέντεγκαρτ για την εκτενή αυτή έκθεση και την ανταλλαγή απόψεων. Ήμουν σχεδόν συζητητή στο παρελθόν για την ένταξη των ε, εναερίων μεταφορών στο σύστημα εμπορία ρήπων και συνειδητά να ενταχθεί αυτό κατά την βούληση τότε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, υπήρξαν ε, προβλήματα τότε, αλλά κάποιος πρέπει να αναλάβει αυτό το ρόλο. Δηλαδή, για τις ε, αφήξεις και αναχωρήσεις που πρέπει να εντάσσονται σε σχέση με την Ευρώπη ως αφετηρία ή ως προορισμό, να εντάσσονται στην εμπορία ρήπων. Και το Σαββατοκύριακο είχαμε και την 7η ναυτιλιακή διάσκεψη στην Ομοσπονδιακή Γερμανία με την Ομοσπονδιακή Καγκελάριο Μέρκελ και είχαμε και σεμινάρια για το περιβάλλον και το κλίμα. Και είμαι ευγνώμων για την δήλωση που <clears throat> στο τέλος του έτους λέει <clears throat> ότι θα υπάρξει νομοθετικό έργο. Οξύδια του αζότου. Για τις εκπομπές οξυδίων του αζότου είχαμε μια ερώτηση που είχε υποβληθεί. Χαιρόμαστε που συμπεριλαμβάνεται και αυτό. Για τις εκπομπές ρήπων τα οξύδια του αζότου είναι ε, μια σημαντική συνιστόσα. Η αποτελεσματικότητα είναι που μετράει. Μια συνολική προσέγγιση μέσω των τομεακών προσεγγίσεων στον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα να κοιτάξουμε ένα όχημα. Τι είναι αυτά που εκπέμπει ο ρήπους για το θέμα των ηλεκτροκινητήρων. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παράγεται αυτή η ενέργεια. Αλλά θα πρέπει συνολικά να δούμε πώς θα παράγεται ένα όχημα. Δηλαδή από τον χάλιβα ή το αλουμίνιο που θα το ε, ε, δημιουργεί μέχρι και την ε, θα έλεγα μέχρι τα παλιοσίδερα που θα είναι το παλαιό αυτοκίνητο που θα ε, οδηγείται στην, το πω έτσι, στην, ε, στον αφοπλισμό, ε, στην απόσυρση από την κυκλοφορία. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα και σε σχέση με έναν κινητήρα που χρησιμοποιεί περισσότερο, περισσότερη ενέργεια Πρέπει να δούμε και για τον κύκλο ζωής του ότι χρειάζεται σημαντικά μεγαλύτερο, μεγαλύτερη ενέργεια. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις βιομηχανίες, ε, στα εργοστάσια που παράγουν ε, καθαρά οχήματα να έχουμε και την προσέγγιση πώς παράγονται αυτά και με ποια μηχανήματα και τεχνολογία. Επόμενος αγορητής παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Κυρία Επίτροπε, άκουσα προσεκτικά αυτά που είπατε στην αρχή της παρέμβασής σας. Μας τα είχατε ξαναπεί θα έλεγα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης την οποία είχαμε με τον Επίτροπο Ταγιάννη και με σας στην Ιδία εδώ και λίγο καιρό. Θα πρέπει να τεθεί λοιπόν το θέμα των επενδύσεων, των σχετικών με τους ανταγωνιστές μας για τις εκπομπές καυσαερίων που δεν προέρχονται από τον άνθρακα βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες οικονομικές εξελίξεις οι οποίες ε, ε, έχουν αρχίσει να φαίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι υπάρχουν επίσης αντίστοιχες εξελίξεις σε πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς τους ανταγωνιστές μας στην Κίνα και αυτό ισχύει και στον τομέα των εκπομπών μη ανθρακούχων καυσαερίων. Να σας θυμίσω επίσης όταν είχαμε συζητήσει και ψηφίσει την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική υπήρξε μια τροπολογία η οποία έτυχε της υποστήριξης της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου που ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια μελέτη σχετικά με έναν πιθανό μηχανισμό του, του υπολογισμού των, των καυσαερίων από άνθρακα αυτή τη φορά στο εσωτερικό των εθνικών συνόρων. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, θα πρέπει να μελετηθεί έτσι ώστε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών μας. Ευχαριστώ. Κράμερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Έχω κι εγώ ένα ερώτημα για τις αεροπορικές εταιρείες. Πρέπει να δούμε την κατάσταση εκεί πέρα να μην ωρεοποιούμε τα πράγματα, γιατί το θέμα δεν είναι πως έχουμε κράτη-μέλη που δεν είναι ικανοποιημένα και πρέπει να τα πείσουμε, αλλά πλέον έχουμε ε, συγκεκριμένα αντίμετρα. Έχουμε υποθέσεις ε, που πάνε στο ΔΕΚ, έχουμε επίσημη ε, θέση της κινέζικης κυβέρνησης πώς θα επιβάλλει καταναγκαστικά τέλη σε ευρωπαϊκές εταιρείε εάν γίνει κάτι τέτοιο, οπότε πως έχουμε δικαίωμα ε, μισό έτος πριν τεθεί η αυτή νομοθεσία να μάθουμε τι κάνει η Κομισιόν. Είναι σαφές πως θα πρέπει να έχουμε ισοδύναμα μέτρα γιατί βεβαίω δεν μπορούμε να εξαναγκάσουμε τα, τα, τις τρίτες χώρες αν δεν θέλουν. Με ποια κριτήρια λοιπόν αυτά θα οριστούν αυτά τα ισοδύναμα μέτρα να υποθέσουμε πως θα αποδεχτεί ισοδύναμα μέτρα η Κομισιόν που θα ανταποκρίνονται μόνο στο κόστος ε, της Ευρώπης. Αλλιώς θα εξαναγκάσουμε πλέον ε, τις ευρωπαϊκές εταιρείε να επομιστούν κόστος το οποίο δεν θα έχουν οι ανταγωνιστές τους. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν ποια σχέδια έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Γιατί εντάξει, μην ωραιοποιούμε τα βάρματα, Είναι σαφέ πω θα πρέπει να οδηγηθούμε σε αυτά τα ισοδύναμα μέτρα. Ποιε Ποιου όρου θα έχουν λοιπόν αυτά τα ισοδύναμα και πότε μπορούμε να αναμένουμε δημοσιοποίηση. Ευχαριστώ. Dan Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, συχνά έχετε πει και είπατε και σήμερα πως εάν πάμε σε ένα στόχο 30% αντί για 20% ε, θα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και όχι το αντίθετο. Εγώ είμαι πεπισμένος πως αύριο η Επιτροπή μας θα σας στηρίξει σε αυτό. Και μάλλον θα έχουμε και πλειοψηφία στην Ολομέλεια σε ένα μήνα από τώρα. Από το ερώτημά μου είναι σαφές. Τι θα χρειαστεί για να καταθέσετε μια νομοθετική πρόταση. Κάνατε την ανάλυση και λέτε πως είναι σαφ... καλή ιδέα. Έχετε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πότε, πότε θα έχουμε την, την πρόταση για να ξεκινήσουμε. Γιατί εάν ε, είναι να έχουμε το πλεονέκτημα το ότι είμαστε πρωτοπόροι πρέπει να ξεκινήσουμε. Τονίσατε κι εσείς συχνά πως η Κίνα δεν περιμένει και πρέπει κι εμείς να κινηθούμε. Μπορείτε επίσης να μας πείτε ε, κάποια πράγματα για το COP17 στην Νότιο Αφρική. Πού βρισκόμαστε τώρα και ποια είναι η στρατηγική της Ένωσης μέχρι αλλά μπορούμε να, μπορείτε νομίζω να έχετε μια αρχική αξιολόγηση του πού πάνε τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έχουμε άλλους δύο που πανε τα πραγματα ευχαριστω ευχαριστω εχουμε αλλους δυο που ζητουν τον λόγο. Λάουσεν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κάποιες ερωτήσεις προς την κυρία Επίτροπο. Πριν από κάποιες εβδομάδες εσείς από κοινού με τους επιτρόπους για το περιβάλλον και την γεωργία είχατε αναφέρει τον συσχετισμό των θεμάτων περιβάλλοντος, κλίματος. Είναι δυνατόν, διαρωτώ με, όλα αυτά να τα πάρουμε με κάθε σοβαρότητα έτσι, διότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση τόσο γοργά όσο θα έπρεπε όσον αφορά τις ε, εκπομπές ρήπων, όσον αφορά τις αρρώσιμες εκτάσεις και τη δασοκομεία παγκόσμια. Το γεγονός είναι, λένε οι επιστήμονες, ότι αν καταρχήν είχαμε γεωργία παγκόσμια χωρίς ε, άρρωση της γης, χωρίς να οργώνεται η γη, 40 χρόνια θα μπορούσε να ε, ε, δεσμευτεί το διοξίδιο του άνθρακα. Μιλάμε για τεράστια ποσά. Ίσως θα πρέπει να το δούμε αυτό σε μια κλίμακα. Και τώρα υπάρχει αυτό το ζήτημα. Δεν θα έπρεπε να καλλιεργούμε βιοκαύσιμα σε αρρώσιμες εδάφεις που μπορούν να παράξουν τρόφιμα. Είναι επίσης και πάρα πολύ επικίνδυνο αυτά τα απόβλητα όπως τα αποκαλούμε από την γεωργία να καίγονται θα έπρεπε να αποθηκεύονται για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Είναι καλύτερο ξύλο να παίρνει κανείς και αυτό να ε, μετατρέπεται μετά να μπορεί να χρησιμοποιείται σε, ε, στη δημιουργία επίπλων και όχι να υπάρχει αυτή η καύση. Αν χρησιμοποιούσαμε όλη την βιομάζα τότε θα ε, μπορούσαμε να προχωρήσουμε και να ε, σημειώσουμε πρόοδο. Θα μπορούσαμε να ελέγξουμε και τις ε, εκπομπές τρύπων και τα οξύδια του αζότου επιπλέον. Ευχαριστώ. Judith Μακής, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ, Πρόεδρε για την παρουσίασή σας. <laughs> Μια τεχνική ερώτηση. Έχω θέσει το ερώτημα αυτό και μας έχετε ήδη δώσει παλαιότερα μια γραπτή απάντηση. Μια πρώτη απάντηση θα έλεγα. Πότε θα ξεκινήσετε να εφαρμόζετε τα διορθωτικά μέτρα και τις διαδικασίες επί παραβάση εναντίον χωρών που δεν εκπληρούν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τους στόχους του 2020. Στη δική μου χώρα είναι σαφές ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει πει ότι θα προσπαθήσει, θα προσπαθήσει να πετύχει τους συμπεφωνημένους στόχους, αλλά δεν είναι βέβαιοι ότι θα το πετύχουν αυτό. Το ερώτημά μου είναι πότε θα λάβετε διορθωτικά μέτρα. Είπατε στην πρώτη απάντησή σας ότι η διορθωτική δράση θα αναλυφθεί ανάλογα με και σύμφωνα με το άρθρο 7. Ε, ποια είναι αυτή η διορθωτική απάντηση. Αν μια έκθεση ελέγχου, σαν παράδειγμα, δείχνει ότι ένα συγκεκριμένο έτος ένα κράτος μέλος δεν είναι συμβατά αυτά που κάνει με τους στόχους και λέτε εσείς ότι θα ξεκινήσετε ίσως μια διαδικασία αν δεν υπακούσει στην ομοθεσία ένα κράτος μέλος, αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν. Εμείς θα λάβουμε διορθωτικά μέτρα το 2020 όταν δούμε ότι τα κράτη-μέλη δεν θα έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους ή θα ξεκινήσετε την εφαρμογή τέτοιων κυρώσεων ουσιαστικά ενωρίτερα. Ευχαριστώ και τελευταία παρέμβαση η κυρία ευχαριστω και τελευταια παρεμβαση κυρια Βέσλοντ. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ ένα ερώτημα για τις δημόσιες προμήθειες. Αυτή τη στιγμή σας απασχολούν ε, στην Επιτροπή ως Επίτροπος Κλίματος. Τι θα θέλατε να αλλάξετε περισσότερο στους κανόνες περί δημοσίων προμηθειών για να βοηθήσετε αυτούς που θέλουν να έχουν έξυπνες προμήθειες και να εμπλακεί και περισσότερος κόσμος. Ε, τι θα προτείνατε ως προς αυτό. Και έχω και άλλη μία ερώτηση και αυτό αφορά τις χαλιβουργίες και βιομηχανίες αλουμινίου στην Ευρώπη που δεν κολλάνε πάρα πολύ με το σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών γιατί είναι εκτεθειμένοι σε πολύ ανταγωνισμό. Οπότε το ερώτημά μου είναι υπάρχουν συζητήσεις με άλλες χώρες για να έχουμε κάποιες τομεακές συμφωνίες για αυτές τις βιομηχανίες και ποιες είναι αυτές οι χώρες. Μάλιστα, πολλές οι ερωτήσεις και τώρα αναμένουμε τις απαντήσεις σας. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από τέλος. Πράγματι υπάρχει τομεακή συνεργασία. Συζητήσεις, παραδείγματος χάρη με την Κίνα, το προτείναμε αυτό πέρσι τον Απρίλιο και έκτοτε τρεις φορές μια ομάδα της Κομισιόν και μια κινέζικη ομάδα έχουν συναντηθεί υπήρχε, εμείς αφορούσα, το θέμα αφορούσε λοιπόν τις ενεργοβόρες βιομηχανίες για να συνεργαστούμε και διμερώς με κάποιους εταιρείες, όχι μόνο στις διεθνείς Τώρα για το άλλο κομμάτι της ερώτησης, το τι θα ήθελα εγώ να κάνουμε για να έχουμε έτσι, μια κινητοποίηση με τρόπο υπέρ του κλίματος. Είναι σημαντική σήμανση, σωστός μηχανισμός τιμολόγησης, γι' αυτό και η οδηγία φορολόγησης της ενέργειας που είναι πάρα πολύ σημαντική εδώ πέρα και οι πράσινες δημόσιες προμήθειες επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί ο δημόσιος τομέας σε όλα τα κράτη-μέλη έχει τεράστια αγοραστική δύναμη και μπορεί να προωθήσει νέα προϊόντα στην αγορά και να τα κάνει πιο διαθέσιμα, πιο φτηνά για τον απλό πολίτη. Ο κύριος Πρόεδρος ρώτησε για την Κίνα και τους διαφορετικούς τίτλους εκεί πέρα, το τονίσετε πάρα πολύ και τους τίτλους των εφημερίδων βεβαίως, Ματίας Γκρότε και λοιποί. Να πω μόνο πως υποθέτω πως όταν η προηγούμενη Επιτροπή μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισαν να συμπεριλάβουν την αεροπορία στο σύστημα εμπορίας εκπομπών με τον τρόπο που έγινε, δεν ήταν τυχαίο αυτό. Και θα ήταν αφελές να πιστεύουμε πως θα ήταν κάτι το εύκολο. Ναι, βεβαίως υπάρχει τώρα κόσμος που έχει μάθει σε στόχους για το κλίμα, ε, αυτά δεν είναι για μας. Και τώρα η Κίνα λέει γιατί εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Είναι εύκολο να δει κανεί ε, το γιατί του συμφέρει αυτό. Κάποιος ρώτησε τι κάνουμε. Είχαμε συναντήσει με τις αρχές, ε, τις πολιτικές αρχές και με τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, οπότε υπάρχει ένας διάλογος και ίσως προσέξατε πως ε, πριν από λίγες εβδομάδες η Κίνα για πρώτη φορά ε, έκανε μια πρόταση να έχουν το στόχο μείωση για την αεροπορία, ένα 22% σε σχέση με τα συνήθη. Τώρα προσπαθούμε να δούμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή θα είναι ισοδύναμα μέτρα ή κάτι άλλο. Το εξετάζουμε γιατί διαμαρτύρονται αλλά ταυτόχρονα προτείνουν και κάποιες πρωτοβουλίες στον τομέα αυτών. Επίσης, για να ξεκαθαρίσω και κάτι άλλο, φαντάζεστε εμείς να κάνουμε τέτοια νομοθεσία στην Ευρώπη και μόλις να αφισβητήσει κάποιος εκτός Ευρώπης να πούμε «Α, Αχ, όχι, συγγνώμη, πλάκα κάναμε. Ε, δεν είναι τρόπος αυτός να πείσουμε την Κίνα και τους άλλους. Ε, Οπότε δεν θα πρέπει τώρα να αγχωνόμαστε. Υπάρχει λόγος να πούμε πως οι πτήσεις που αναχωρούν και προσγειώνονται στην Ευρώπη θα πρέπει να συνεισφέρουν στον αντίκτυπο που έχουν στο κλίμα. Πήγα στο Χονγκ Κονγκ πρόσφατα και εκεί πέρα έλεγαν γιατί να πληρώνουμε εμεί Και κάποιες αεροπορικές εταιρείε έλεγαν γιατί να πληρώσουμε εμεί. Γιατί ένας επιχειρηματίας από το Χονγκ Κονγκ που μπορεί να πληρώσει το εισιτήριο με την Cathay Pacific να έρθει στο Λονδίνο να μην ε, ενταχθεί στην αρχή ορυπαίνων ε, πληρώνει. Ποια λογική έχει αυτό ενώ ο φοιτητή που πάει στο πανεπιστήμιο για να επισκεφθεί τους γονείς του να πληρώνουν αυτοί. Υπάρχουν κάποιες αρχές εδώ πέρα που πρέπει να ισχύσουν. Ό,τι έγινε έγινε συνειδητά και πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι τώρα και ας αμφισβητούν μερικοί για, επειδή δεν θέλουν να πληρώσουν. Και να τονίσω πως σύμφωνα με τη σύμβαση του Σικάγου ό,τι συμβαίνει στο αεροδρόμιο αναχώρησης ε, εξαρτάται 100% από αυτή τη χώρα. Και βλέπουμε και την απόφαση την τελευταία του ΙΚΑΟ ε, στον Καναδά ε, το φθινόπωρο που είπε πως μπορούμε να έχουμε περιφερειακά συστήματα εμπορίας εκπομπών. Λίντα Μακιούαν και άλλοι ανέφεραν τον παράγοντα Άιλουκ θα ξέρετε φαντάζομαι πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πετύχουμε σωστά αυτό το θέμα. Επίσης να σας πω πως δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό γιατί η επιστήμη ακόμα, η γνώση ως προς αυτό δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ αλλά π.χ. η Λίντα ανέφερε την αρπαγή γη στην Αφρική κτλ. Όλοι ξέρουμε γιατί είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να δούμε αυτό το ζήτημα παρά το ότι είναι δύσκολο. Επίσης αναφέρεται Μπασάικχουτ τη... τα σχιστολιστικά κοινά πετρώματα που περιέχουν ε, πετρελαίο και είδαμε τώρα τα τις επιστημονικές μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί και για να υπάρχει πλήρης ε, διαφάνεια η Κομισιόν οργανώνει μια συνάντηση των ενδιαφερομένων αυτή την Παρασκευή, Παρασκευή 27 για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα ακριβώς της μελέτης αυτής επιστημονικής. Οπότε ξέρετε γιατί πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Βεβαίως, ο Καναδάς δεν είναι ικανοποιημένος όπως ε, φαντάζεστε, αλλά ξέρω πως ε, και οι βουλευτές ε, είχαν προσκληθεί την Παρασκευή. Οπότε προχωράμε. Μετά, το ερώτημα για την κοινή πολιτική και την πολιτική αλίας. Ναι, αυτή τη στιγμή συζητάμε αρχές εντό τη Κομισιόν και τέτοια ζητήματα, αλλά είμαστε ακόμη στην πρώτη ε, φάση. Αλλά όπως επίσης αναφέρθηκε, ε, γράψαμε και μια κοινή επιστολή, η Επίτροπη Ποτότσνικ, ε, Τσόλος και εγώ, προς κάποιους υπουργούς για την κοινή γεωργική πολιτική για να δούμε για για να παρουσιάσουμε το γιατί πρέπει να έχουμε πιο πράσινη κοινή πολιτική. Βεβαίω το συζητούσαμε αυτό σχέση με τον... Πώ μπορούμε να προσθέσουμε πρόσθετη αξία σε σχέση και με τι επιδοτήσει για τη γεωργική πολιτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί το θέμα των επιδοτήσεων. Μπορεί να πρασινίσει η Γεωργία και όχι μόνο στον πρώτο πυλώνα το πρασίνισμα, αλλά και στον δεύτερο πυλώνα. Πώς μπορεί τεχνολογία και συναφείς δράσεις. Έχουμε ουσιώδεις συζητήσεις από αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όταν θα υποβληθούν οι προτάσεις μας και πριν από την 1η Ιουλίου, μετά θα είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να τοποθετηθεί και να διαδραματίσει ρόλο επ' αυτόν. Μπορούμε να έχουμε πολύ μεγάλη πρόσθετη αξία σε σχέση με την ΚΑΠ. Και όσον αφορά τον οδικό χάρτη, όπως γνωρίζετε, που σημείωσε τι κάθε κράτος έχει από πλευρά σχεδίων για το ενεργειακό μείγμα όσον αφορά και την ε, ε, πυρηνική εκμετάλλευση. Αυτό αποτελεί ένα, ε, μια συνιστόσα. Η Γερμανία έχει ένα, ένα ξεχωριστό ρόλο να διαδραματίσει εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα μετά ε, την Φουκουσίμα να το αναγνωρίσουμε, να συζητήσουμε το θέμα της αποδοτικότητας ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας. Και 25 ο οδικός ε, χάρτης για την ενέργεια αυτό προσκαλεί να γίνει. Και σε σχέση με αυτό τον οδικό χάρτη είχαμε ενδεικτικούς στόχους που πρέπει να καταλήξουμε στο 2030 ε, με τις εκπομπές τρύπων. Είναι τώρα η χρονική στιγμή να αρχίσουμε έγκαιρα να συζητήσουμε το θέμα στόχου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπό διαφορετικό πρίσμα μπορεί να προσεγγίσει κανείς αυτά τα θέματα και σε σχέση με το οδικό χάρτη του 2005 είναι μια λογική συζήτηση που πρέπει να διεξαχθεί αυτή προηγούμενα μετά την Φουκουσίμα να μην ε, ε καταλήξουμε, ε, κολλήσουμε περισσότερο στα ορυκτά καύσιμα και ή καταστήσουμε υπερβολικά δαπανηρό να έχουμε, ας το πω έτσι, μια ε, με λιγότερους ε, ενεργειακή χρήση. Αναφέρθηκε από τον Chris τι θα γίνει σε σχέση με το 2050. Το επόμενο βήμα θα είναι η συζήτηση αυτών. Το Συμβούλιο θα πρέπει να, να αποφασίσει για την αποδοτικότητα της ενέργειας και το πρόγραμμα δράσης για το ποσοστό των δημόσιων κτηρίων που θα πρέπει να, ε, να, προσαρμόζονται σε σχέση με την αποδοτικότερη χρήση ενέργειας ε, και πρέπει αυτά να συζητηθούν στο Συμβούλιο και να προαχθούν και μετά από την ανακοίνωση που έγινε το 2010 ξεκινήσαμε μια ανάλυση ανακράτος μέλος των πραγμάτων και θα υποβληθεί αυτή η ανάλυση πριν από το, τις θερινές διακοπές και έτσι θα είμαστε έτοιμοι για κάποιους μήνες μετά στη συνέχεια κατά τέλη του έτους με το Συμβούλιο να συζητήσουμε τι όλα αυτά συνεπάγονται, ποιες επιπτώσεις έχουν όλα αυτά για τα επιμέρους κράτη-μέλη, ποια προσέγγιση ακολουθούν τα κράτη-μέλη. Αυτά είναι τα αμεσότερα πράγματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από πλευρά μας με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω έχω ήδη απαντήσει στην παρέμβαση του Ματίας Ρόντε και για τις εναρίες μεταφορές. Ρώτησε επίσης και για τον χρόνο, κύκλο ζωής ε, και την αξιολόγηση των αυτοκινήτων, των οχημάτων. Πρέπει να υπάρξει ε, αυτή η ε, διάσταση, αυτή η συνιστόσα. Προετοιμάζει το, πρόγραμμα, το νομοθετικό πρόγραμμα για την αποδοτικότητα ενέργειας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εξεταστεί, και η, θα εξεταστεί αποδοτικότητα και στα μέτρα παραγωγής. Θα πρέπει εδώ να δούμε και το θέμα της ίσως επικαιροποίησης της σημερινής νομοθεσίας αλλά θα πρέπει να παραμείνουμε μέσα στους στόχους που, στους στόχους που έχουμε θέσει. Ρωτήσατε όταν θα έχουμε τώρα μια πρόταση που θα υποβληθεί στα κράτη-μέλη με ανάλυση ανα, κράτος μέλος προς κράτος μέλος μετά από μερικούς μήνες όπως προανέφερα θα πρέπει να δούμε με τα κράτη-μέλη ποιο είναι το δυναμικό τους, ποιες είναι οι αντιδράσεις τους. Ξέρω και από κάποια κράτη-μέλη και καινούρια κράτη-μέλη σε σχέση με τους στόχους ε, για το 2020 ε, χώρια που ε, προσεγγίζουν μακροπρόθεσμους, πιο μακροπρόθεσμους στόχους. Είναι σε σχέση με τον προϋπολογισμό κέρια σημασία αυτό. Να δοθεί το μήνυμα στα κράτη-μέλη ότι θα υπάρξει βοήθεια όταν θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο φιλόδοξοι, τότε μπορούμε να πετύχουμε πρόσθετη αξία και υποστήριξη από τα κονδύλια του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτέ τι προσπάθειε. Αυτό είναι τμήμα τη συζήτηση που διεξάγεται τώρα. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική έκβαση μέχρι τον Ιούλιο, αλλά είναι ουσιώδη αυτά τα θέματα. Μετά ρωτήσατε για τα θέματα ε, που ε, ε, αφορούν την μείωση και όσον αφορά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μεριμνήσουμε ότι θα υπάρξουν και άλλα θετικά αποτελέσματα στη σε σχέση με τα πιο δυσχερή ζητήματα. Είμαστε πρόθυμοι να δούμε υπό την, ε, διάδοχο, υπό την ε, Επιτροπή και το έργο που θα ακολουθήσει πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν. Αυτά όταν η Ιαπωνία, η Ρωσία και οι άλλοι, όταν έχουν αντιστάσεις και λένε ότι δεν είναι πρόθυμοι να αναλάβουν δεύτερες ε, πρόσθετες δεσμεύσεις. Αν το κάναμε εμείς πώς θα βοηθούσε αυτό. Θα βοηθούσε η οικογένεια εκείνων που θα ήταν υπέρ μιας δεσμευτικής συμφωνίας να αυξηθεί, να επεκταθεί ή θα αποδυναμωνόμαστε γιατί θα συρρυκνωνόταν η οικογένειά μας αυτή. Αυτή είναι η οικογενεια μα αυτη αυτη ειναι η συζητηση που διεξάγεται τώρα για αυτά τα θέματα. Προσπαθούμε να προωθήσουμε αυτά και στις ε, συζητήσει στις Βρυξέλλε μετά το ε, Πάσχα τα θέματα αυτά σημειώνουν με βραδείς ρυθμούς ε, πρόοδο, ίσως υπερβολικά βραδεί ρυθμούς. Προσπαθούμε να στείλουμε σαφή μηνύματα στους Νοτιοαφρικανούς ότι είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους βοηθήσουμε. Αλλά πρέπει να υπάρχει σαφή στοχοθέτηση. Θα έχουμε διαπραγματεύσει σύντομα και θα έχουμε και γύρω στις αρχές Ιουλίου ε, τη συνάντηση με τους υπουργούς θα προσπαθήσουμε να σημειωθεί ουσιώδης πρόοδος γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Θα έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε ούτως ή άλλως. Αυτά πρόεδρε εν συνόψη και σε σχέση με το ερώτημα πότε θα ξεκινήσουμε με τις κυρώσεις και τις, ε, ε, την, την τιμωρία των, των παραβάσεων και παραβιάσεων θα υπάρχουν ε, οι, ε, οι μετρήσεις ε, που θα οδηγούν στις κυρώσεις να θα αξιολογούμε αν τα κράτη-μέλη συμμορφώνονται ή όχι και τότε εν δυνάμει θα μπορούμε από το 2013 σε αιτήσια βάση να προσφεύγουμε εις βάρος των κρατών που δεν θα ευθυγραμμίζονται και δεν θα συμμορφούνται. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ για αυτές τις απαντήσεις, κυρία Επίτροπε. Ήταν πραγματικά ουσιώδεις αυτές ε, οι ε, παρατηρήσεις. Κάνουμε το καλύτερο ότι περνάει από το χέρι μας να προαγάγουμε αυτά τα θέματα, κυρίως σε σχέση με τα κράτη-μέλη βέβαια. Να ενθαρρύνουμε, να προτρέψουμε περισσότερο τα κράτη-μέλη, να μην εφησυχάζουν και ιδιαίτερα εκείνοι να υποστηριχθούν, εκείνα τα κράτη-μέλη που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο επιδόσεων, ώστε να είναι προπομπός πρωτοπόρος η Ευρώπη και να δίνει το παράδειγμα σε άλλους ε, που θα ακολουθήσουν αυτή την πορεία. Και καθοδόν προς τον Τέρμπαν θα έχουμε και άλλες συζητήσεις. Θα δούμε ποια θα είναι η συγκεκριμένη θέση που θα αποκρισταλωθεί για μας. Όταν λέμε για το Κιώτο έχουμε και το θέμα της ε, Νορβηγίας και της Ελβετίας πώς μπορούν να βοηθήσουν ε, και το θέμα είναι ότι πιστεύουμε ότι ο μηχανισμός του Κιώτο πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω, να μεταξελιχθεί και η Ευρώπη να μπορέσει να, εντα, να προωθήσει αυτά τα θέματα έναντι εκείνων που δεν θέλουν να συμμετάσχουν. Κάθε επιτυχία σας εύχομαι και θα συναντηθούμε και με την επόμενη εκδήλωση, στην επόμενη ευκαιρία. Ευχαριστώ. So, Οπότε συνεχίζουμε κανονικά. Είπαμε ήδη καλημέρα. Εμείς είχαμε ζητήσει λοιπόν αυτήν την συζήτηση οι συντονιστές, δηλαδή μια ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο και καλωσορίζω τον πρόεδρο τον κύριο Φιλίπ Μάιστατ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία θέλει η πολιτική πρέπει να χρηματοδοτηθούν και ένα μέσο της Ευρώπης είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Βεβαίως ε, μας ενδιαφέρει να ακούσουμε το πόσο στηρίζεται αυτούς τους πολιτικούς στόχους και τα προγράμματα γιατί δεν έχουμε πάρα πολλά μέσα. Είστε νομίζω το πιο μεγάλο και επιφανή μέσο τη ε, ένωση για την προστασία του κλίματο στην Ευρώπη και εκτός Ένωση. σε άλλες ε, υπήρους. Θα σας δώσω λοιπόν όμως τον λόγο και αναμένουμε αυτό το οποίο θα μας πείτε και ευχαριστώ που ήρθατε. Merci, Monsieur le Président. Et Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα να ομιλήσω εδώ. Αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημιουργήθηκε από τη συνθήκη της Ρώμης για να υποστηρίξει τους στόχους αυτού που ονομάζαμε κάποτε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, αλλά σήμερα τους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταπολέμηση των κλιματολογικών συνεπειών είναι μία από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι λογικό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κληθεί, να συνεισφέρει και αυτή από πλευράς της. Δεν θα ήθελα να επιμείνω εδώ για την σημασία που έχει η καταπολέμηση των συνεπειών των αλλαγών αυτών. Για να πετύχουμε όμως τους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει αυξημένη ανάγκη επενδύσεων. Η Επίτροπος Χέλντεγκαρντ, της οποίας θαυμάζω την αποφασιστικότητα, το είπε ήδη, και θεώρησε μάλιστα ότι οι ανάγκες των επενδύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνουν περίπου στα 270 δις κατέτος για τα επόμενα 40 χρόνια. Ε, πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό βέβαια και όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε θα πρέπει οι επενδύσεις αυτές να μπορέσουν να τύχουν χρηματοδότησης και αυτό ε, σε κάποια πλαίσια όπου τα δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται υποπίεση τα μέσα δηλαδή ε, δημοσίων χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων είναι σχετικά περιορισμένα και παραμένουν περιορισμένα. Από την άλλη, οι τραπεζικές χρηματοδοτήσεις για τέτοιου είδους επενδύσεις, οι οποίες απαιτούνται να γίνουν σε μακροπρόθεσμη βάση, είναι σαφές ότι ο γερμανοπιστωτικός, ο τραπεζοπιστωτικός τομέας θα επιβραδύνει την παρέμβασή του λόγω ακριβώς των κανόνων Βασιλεία 3 και όλοι εν πάση περιπτώσει ελπίζουν ότι δεν θα περιορίσουν ιδιαίτερα οι νέοι αυτοί κανόνες την ικανότητα του πιστοτικού τομέα να προχωρά σε μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις. Είναι σαφές λοιπόν ότι κάτω από τις συνθήκες αυτές στρεφόμεθα προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σας είπα ότι είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε, να συνεισφέρουμε Βέβαια εμείς δεν μπορούμε να προσφέρουμε την μαγική λύση, έχουμε και εμείς περιορισμούς, ιδιαίτερα περιορισμούς σε επίπεδο κεφαλαίων, γιατί όπως και όλες οι τράπεζες πρέπει εμείς να σεβαστούμε τους, ε, τη σχέση ε, των επενδυωμένων κεφαλαίων με ε, τους σταθμισμένα κεφάλαια και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα τελειώσω εδώ, είναι χρήσιμο να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους που συνδυάζουν ε, τα δημοσιονομικά μέσα της Ένωσης με τα μέσα της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που θα λειτουργήσουν σαν μοχλός που θα διευκολύνει και τις δύο πλευρές. Ε, να παρουσιάσω τώρα πάρα πολύ σύντομα αυτά τα οποία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κάνει σήμερα ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Νομίζω ότι σας έχουν ήδη διανύμει κάποιους πίνακες οι οποίοι δείχνουν καταρχάς ότι έχουμε αυξήσει ε, σημαντικά τις χρηματοδοτήσεις μας στον τομέα της ενέργειας. Περάσαμε από 4 δις το 2006 σε 18 δις το 2010, μια ουσιαστική αύξηση δηλαδή της χρηματοδότησης στον τομέα της ενέργειας, όπως βλέπετε στον πίνακα που έχετε, εδώ βλέπετε τι ακριβώς κάνουμε. Το άνω τμήμα του πίνακα, σαν ανοιχτό πράσινο, είναι οι επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Όλοι αναγνωρίζουν ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να μειώσει κανείς το ενεργειακό κόστος, να καταναλώνει δηλαδή λιγότερη ενέργεια. Και αυτή είναι μια βασική λοιπόν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Notamment grâce à un programme qui a été lancé avec euh, la, Commission et qui est le λοιπόν, και υπάρχει και το πρόγραμμα Ελένα, το οποίο έχει σαν στόχο να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να προετοιμάζουν κάποια προγράμματα βελτίωσης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Είναι ένα πρόγραμμα, θα έλεγα πρόσφατο, Ήδη έχουμε βοηθήσει σε τεχνικό επίπεδο 11 προσπάθειες δήμων και κοινοτήτων για την εφαρμογή τέτοιου είδους προγραμμάτων. 20 εκατομμύρια τεχνικής βοήθειας που υποστηρίζει επενδύσεις ενός δις 600 εκατομμυρίων. Ένα παράδειγμα. Το τι έχουμε κάνει με την επαρχία του Μιλάνου στην Ιταλία το 2006 η επαρχία αποφάσισε να κάνει ε, ενεργειακούς ελέγχους αλλά λόγω έλλειψης χρημάτων και ε, λόγω ελλείψεων τεχνικών δεν προχωρήσανε. Αλλά χάρη στο πρόγραμμα Ελένα μπόρεσαν ε, επί τη βάση των ελέγχων που έγιναν να κάνουν βήματα, να ομαδοποιήσουν τα προγράμματα, να ομαδοποιήσουν την αγορά εξοπλισμών να δημιουργήσουν ε, συμβόλαια τύπους και έτσι μπόρεσε η τράπεζα να δώσει 65 εκατομμύρια για την ανακαίνιση των δημοσίων σχολείων σε 30 σχολεία της επαρχίας του Μιλάνου. Αυτού του είδους τα προγράμματα, εφόσον εκτελούνται σωστά, είναι ακριβώς υποδειγματικά θα έλεγα για την χρήση τους και σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Να αναφερθώ επίσης στο πρόγραμμα Jessica, το οποίο χρησιμοποιεί χρήματα των διαφορετικών ταμείων. Στην Λιθουανία η Jessica σαν παράδειγμα έχει χρηματοδοτήσει μακροπρόθεσμα την αποκατάσταση ε, πολυκατοικιών παλαιού τύπου. Και τέλος, ε, ένα άλλο τομέα, τον οποίο γνωρίζετε, βρισκόμαστε στην τελευταία φάση της δημιουργίας ενός ειδικού ταμείου, το οποίο θα προσπαθήσει να βοηθήσει στην σωστή χρηματοδότηση των 146 εκατομμυρίων που περίσεψαν από το πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης, το τόσο γνωστό. Αυτός είναι ένας τομέας λοιπόν βασικός για μας στο μέλλον. Πέρυσι δανείσαμε 230 εκατομμύρια στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα αυτό της ενέργειας και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε και να αυξήσουμε τις χρηματοδοτήσεις μας. Πάντα στον ίδιο πίνακα. Βλέπετε με σκούρο κιανό χρώμα τις χρηματοδοτήσεις μας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ εντασσόμεθα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2009 που παρακινεί τα κράτη-μέλη να στηρίξουν την ανάπτυξη των ε, εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Είναι απαραίτητο να γίνει γιατί όπως ξέρετε υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά στο κόστος της παραγωγής ενέργειας ανάμεσα στον παραδοσιακό τρόπο και στον τρόπο παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές Βέβαια βλέπει κανείς ότι η διαφορά μειούται λόγω των οικονομιών κλίμακας και της προόδου της τεχνολογίας και βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος. Παρ' όλα αυτά για κάποιο χρονικό διάστημα αυτοί οι μηχανισμοί στήριξης πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν. Πρέπει να αποφύγουμε βέβαια <clears throat> αναδρομικά μέτρα γιατί σε περιπτώσεις ε, δημοσιονομικής σύσφυξης θα έλεγα είναι θα έλεγα εύκολο να εγκαταλείψει κανείς τέτοιου είδους προσπάθειες γιατί αυτό δεν θα ήταν καλό, θα δημιουργήσει αβεβαιότητα στους επενδυτές οι οποίοι καλούνται από την άλλη να επενδύσουν περισσότερα. Στον τομέα των εναλλακτικών πηγών ενισχύσαμε τις παρεμβάσεις μας από 500 εκατομμύρια το 2006 σε 6 500 εκατομμύρια το 2010. Δεκαπλασιάσαμε δηλαδή την προσπάθειά μας. Και ακριβώς στα πλαίσια της δημοσιονομικής κρίσης όλα, η τράπεζά μας έπαιξε αποφασιστικό ρόλο για ορισμένα προγράμματα. Λειτουργήσαμε σαν α, α, κομβικός επενδυτής, cornerstone investor και για τη Βόρεια Θάλασσα ξεκίνησε το πρόγραμμα του 2009 λόγω ακριβώς της έλλειψης οικονομικής στήριξης. Είχαν αποσυρθεί κάποιοι επενδυτές. Αυτές οι ε, ε, εν μέσω της θαλάσσης αιωλικές εγκαταστάσεις και η τράπεζά μας έδωσε 300 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα το οποίο του επέτρεψε να αναδιοργανωθεί και γι' αυτό ακριβώς πήραμε και το βραβείο του καλύτερου δανειστή για τις ανανεώσιμες πηγές, λόγω ακριβώς αυτής της παρέμβασής μας η οποία έσωσε την προσπάθεια αυτή, του πρόγραμμα αυτό. Μια άλλη προσπάθεια είναι το Μοντεντικάστρο στην Ιταλία. Γιατί εκεί η παρέμβαση της τράπεζάς μας με 100 εκατομμύρια σε δευτερεύοντα δάνεια που επέτρεψε ε, στον εργολάβο να εκδώσει ακριβώς ομολογίες ε, τις οποίες πούλησε σε ιδιώτες ε, επενδυτές. Ε, γιατί ακριβώς λόγω της παρέμβασής μας κατέστησαν ενδιαφέρουσες και συμφέρουσες οι ομολογίες αυτές. Να αναφέρω επίσης τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών, αυτά που κάνουμε σε ορισμένες περιφέρειες, σε γαλλικές ας πούμε, αρκετές γαλλικές περιφέρειες, στο Νότο, στο, στο Ρουσιγιόν, στο Πουατού Σαρόντ, προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε κάποιες μικρές, ε, ε, κάποιες μικρές προσπάθειες στον τομέα της αηφορίας. Εμείς φυσικά δεν μπορούμε να είμαστε σε επαφή με πολλούς δανειζομένους μικρής εμβέλειας. Περνάμε από τοπικές αρχές ή οργανώσεις οι οποίες καθορίζουν τα κριτήρια επί τη βάση των οποίων εμείς θα χρηματοδοτήσουμε ε, κάποιες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές. Δεν έχω κάτι άλλο να πω στον τομέα της ενέργειας. Να πω επίσης ότι δεν χρηματοδοτούμε μόνο ε, τις τεχνολογίες οι οποίες ήδη έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά χρηματοδοτούμε και αυτό είναι αντικείμενο μια συμφωνίας θα έλεγα στην οποία έχουμε καταλήξει κάποιες αναδιόμενες μορφές ενέργειας όπως πιλωτικά προγράμματα, προγράμματα επίδειξης. Ε, les, les premières expériences euh, d'énergie solaire avec euh, concentration, euh, c'est le cas de, de, de plusieurs projets en Espagne. J'ajoute enfin que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 το 2007 έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά κριτήρια, από το 2007 χρησιμοποιήθηκαν πολλά κριτήρια για την χρηματοδότηση μονάδων που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα. Θα πρέπει καταρχάς να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Δεν μπορούμε δηλαδή να χρηματοδοτήσουμε εγκαταστάσεις που αυξάνουν την παραγωγή ενέργειας αυτού του τύπου. Δεύτερη προϋπόθεση. Θα πρέπει οι νέες επενδύσεις να βοηθήσουν σε μία μείωση 20% ε, της συνολικής χρήσης, ε, να είναι σε ένα πλαίσιο που μειούται η συνολική χρήση του άνθρακα. Θα πρέπει να προσφεύγουν στις βέλτιστες δυνατές τεχνολογίες και θα πρέπει επίσης οι εγκαταστάσεις αυτές να είναι carbon capture ready, δηλαδή η σχεδίαση αυτών των νέων μονάδων να είναι απόλυτα συμβατή και να χρησιμοποιεί την τεχνολογία ε, ε, ε, περιορισμού και αποθήκευσης του διοξιδίου όταν αυτό παραχθεί. Σε σχέση με τα αιτήματα λοιπόν τα πολλά τα οποία πήραμε για χρηματοδότηση ε, μόνο 23 αιτήματα εξετάσαμε προσεκτικότερα, τα υπόλοιπα απερίφθησαν και τα τελευταία χρόνια χρηματοδοτήσαμε μόνο τρεις μονάδες. Τρεις μονάδες οι οποίες ε, ε, πληρούν τα κριτήρια τα οποία είχαμε θέσει. Και έχουμε φυσικά την πρόθεση να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, εννοείται επίσης ότι δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα εφόσον υπάρχει φυσικά η προ, εκ των προτέρων συμφωνία της Επιτροπής. Είμαστε το μόνο χρηματοδοτικό σώμα που δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει κανένα πρόγραμμα αν δεν έχουμε λάβει από πριν την σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια μιας συνεννόησης όλων των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά κύριε Πρόεδρε ήθελα να σας πω. Θα ήθελα κλείνοντας να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στην, στην ε, χρησιμότητα μεικτών μορφών χρηματοδότησης ανάμεσα στον, στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Γιατί αυτό. Όταν χρησιμοποιεί κανείς τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραδοσιακά ε, χρησιμοποιείται στο παρελθόν σαν επιδοτήσεις, άπαξ, αν αντί να χρησιμοποιηθούν σαν επιδοτήσεις, συνδυαστούν με τους πόρους της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας θα λειτουργήσει σαν μοχλός ε, για την επιτυχία των επενδύσεων αυτών και από πλευρά μα, αν μπορούμε να συνδυάσουμε τις δικές μας παρεμβάσει με παρεμβάσεις του κοινοτικού προπολογισμού. Ε, υπάρχει μια ελάφρυνση των ε, ετοιμάτων ε, και της ζήτηση κεφαλαίων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα μέσο που λειτουργεί εδώ και κάποια χρόνια, το Risk Sharing Finance Facility για την έρευνα και την καινοτομία. Αυτό το μέσο ε, μοιράζεται θα έλεγα ανάμεσα, ο κίνδυνος ανάμεσα στον προϋπολογισμό και την τράπεζά μας. Με 370 εκατομμύρια του κοινοτικού προϋπολογισμού πριν μερικούς μήνες δόθηκε η δυνατότητα στην τράπεζά μας να δώσει δάνεια 6 δις ε, που οδήγησε σε συνολικές χρηματοδοτήσεις 16 δις. Βλέπετε λοιπόν αυτή την λειτουργία μοχλού που ανέφερα. 300 ε, εκατομμύρια από τη μία φτάνουν σε 16 δις από την άλλη. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι μια αμοιβαία διευκόλυνση. Αν δεν είχαμε αυτή την δυνατότητα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, τότε θα έπρεπε να αφιερώσουμε, να σκλαβώσουμε σε εισαγωγικά στην επένδυση αυτή πολύ περισσότερα μεγαλύτερα ποσά. Μας επιτρέπει λοιπόν η αποκοινού χρηματοδότηση να καταλήξουμε σε μια συνολική επένδυση πολύ υψηλότερη. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε κάθε συμφέρον αναζήτησης αποτελεσματικών μορφών χρηματοδότησης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ κύριε Μεστάτ. Είχε πολύ ενδιαφέρον το να σας ακούσει κανείς εσάς και τα προγράμματά σας. Και θα χρησιμοποιήσω τα γερμανικά που είναι πιο εύκολα για μένα. Λοιπόν, ερωτώντας ε, για άλλη μια φορά το τελευταίο σημείο το οποίο αναφέρατε, συνδυασμός κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με τα ποσά που παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πού υπάρχουν κάποια όρια, τι πρέπει να κάνουμε για να συνδυάζονται περισσότερο αυτά τα κονδύλια. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Γι' αυτό το Ελένα που προαναφέρατε από ό,τι κατάλαβα είναι κονδύλια για την ενδυνάμωση και ανάπτυξη του δυναμικού, για την απόκτηση τεχνογνωσίας, ε, για βέλτιστη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Είναι πολύ αναγκαίο να γίνεται αυτό. Σε όλες τις χώρες έχουμε ανάγκη στο κοινοτικό επίπεδο τέτοιων προγραμμάτων και σχεδίων ενεργειακών που θα καταρτίζονται. Οι προοπτικές αυτού του προγράμματος Ελένα στην επέκταση αυτή και ενδυνάμωση ποιε είναι και με ευχάριστα. Ίσως θα αναμένατε επικρίσεις για το ότι 10% κονδύλια διαθέτεται για πετρέλαιο και άνθρακα. Εγώ θα έλεγα και θα σκεφτόμουν ότι είναι θα ήταν πολύ περισσότερα. Τώρα 15 στο φυσικό αέριο και να δούμε ότι αυτές τις στρατηγικές που ακολουθείτε εσείς ε, που είναι ε, ας το πω έτσι, αναγκαίες. Εκπλήσωμαι ευχάριστα από αυτό που είπατε και τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο ποσοστό θα ε, απαλληφθεί και θα υπάρχουν ε, ανάγκες ε, μετατροπής ούτως ή άλλως. Έχουμε αρκετούς συναδέλφους που ζητούν τον λόγο. Chris Davis πρώτος, παρακαλώ. Well, my points really. Ναι, τα, και τα δύο σημεία που έχω να πω αφορούν τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και το NER 300. Βεβαίως ε, εξαρτάστε εσείς από την ε, Κομισιόν η οποία θα πρέπει να δώσει άδειες πριν ε, μπορέσετε να αποκτήσετε μια αξία αγοράς. Αλλά όταν συμβεί αυτό έχει κάποια ευελιξία η τράπεζα για την πώληση αυτών των αδειών για να υπάρχει το μάξιμο ποσό διαθέσιμο για δέσμευση και αποθήκευση και ανανεώσιμες. Ε, Προφανώ υποθέτουμε πω καθώ ανακάμπτει η οικονομία η τιμή του άνθρακα θα ανέβει και οι άδειε θα γίνουν πιο ακριβές και πιο πολύτιμέ. Δεύτερον, για τον άνθρακα, ναι, ενδιαφέροντα τα στοιχεία πω λίγε και επενδύσεις κατευθύνονται εκεί πέρα, αλλά αναφερθήκατε σε απέτηση να είναι κάποια πράγματα έτοιμα για δέσμευση και αποθήκευση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει να αφήνουμε ξέρω, κάποιο χώρο σε ένα σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για να βάλουμε ε, κάποια μηχανήματα, αλλά και για να αποδείξουν πως υπάρχει κάποιος χώρος αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα και δεδομένου του ότι δεν έχει μεταφερθεί καν στην εθνική νομοθεσία των περισσότερων κρατών κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό και πώς μπορεί να δικαιολογηθεί η επένδυση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Καθλήν. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μάισταρ, δύο θέματα, ένα γενικό και ένα έτσι κάπως ε, που αφορά την ε, αλλαγή πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να φροντίσουμε να επιτύχουμε όλους τους στόχους. Όμως οι αριθμοί του Bankwatch Network μας λένε πως έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Εάν δούμε το τι έγινε μεταξύ 2001 και 2008, το τι δάνεια έδωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, φαίνεται πως πήγαν 18 δισεκατομμύρια σε ορυκτές πηγές ε, ενέργειας. Εντάξει. Λογικά αυτά τα οποία λέτε, αλλά δεν νομίζω να αλλάζει η τάση η οποία εδώ πέρα υπάρχει. Δηλαδή έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη για μεγαλύτερο ποσοστό ανανεώσιμο. Πώς βλέπετε λοιπόν το μέλλον και πώς σκοπεύετε να αλλάξει αυτή η τάση όπως σας είπα. Και μιλάω βεβαίως ε, πρόθεσμα και όσο το δυνατόν πιο <coughs> σύντομα να επενδύεται μόνο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεύτερον, να αναφέρουμε το εξής. Ε, υπάρχουν κάποιοι βουλευτές εδώ μέσα που ε, δίθυναν μία επιστολή για το ρηχείο χαλκού Μομπάνη στην Ζάμπια που αποτελεί ένα υπόδειγμα του τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον και του τι δεν πάει καλά με τις επενδύσεις Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το 2005 εάν δεν κάνω λάθος, ε, έδωσε 48 εκατομμύρια ευρώ η τράπεζα, τα οποία τα συνέδεσε με κάποια σημαντικά κριτήρια που σχετίζονται με το περιβάλλον και τα κοινωνικά ζητήματα. Έπρεπε δηλαδή η εκμετάλλευση του ορυχείου να ωφελήσει ε, το περιβάλλον, ωραία πράγματα δηλαδή, αλλά από ό,τι φαίνεται συνέβη το αντίθετο, δηλαδή το αποτέλεσμα ήταν να επιδεινωθεί το περιβάλλον και να μην μιλήσουμε για τις συνθήκες ζωής ε, των ανθρώπων. και ε, Επιπλέον φαίνεται πως κάποια από τα λεφτά πήγαν ε, για φοροαποφυγή στην Ζάμπια. Και πρόκειται άρα για παράνομη χρήση. Και έρχομαι στις δύο επόμενες ερωτήσεις. Η τράπεζά σας είναι σε θέση να τηρήσει αυτά τα οποία θέτει η ίδια ως όρους όσον αφορά κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και να δει πως πραγματικά υπάρχει μια συνέχεια και μια παρακολούθηση αυτών των πραγμάτων όπως π.χ. για το ρηχείο Μομπάνι στην Ζάμπη αλλά και για τα πάρα πολλά έργα τα οποία χρηματοδοτεί. Ευχαριστώ. Ο από την κάθε προηγούμενα διατυπώθηκε και έτσι αποσύρω την παρέμβασή μου. Πολύ καλά, εξαιρετικά. Λίντα Μακέβεν, παρακαλώ. Um, Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις ε, για την συλλογή και αποθήκευση άνθρακα. Υπάρχει κάποια ανησυχία ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν έχει όλο το δυναμικό για να αξιολογήσει τέτοια προγράμματα έγκαιρα. Μπορείτε να μας πείτε, βρίσκεστε στη σωστή, ας το πω έτσι, πορεία, ώστε έγκαιρα να αξιολογείτε, διότι πρόκειται για επενδύσεις μακροπρόθεσμες και οι επενδυτές πρέπει να ξέρουν τι θα κάνουν με τα κονδυλιά τους. Ένα δεύτερο θέμα είναι αρκετά τεχνικό φύση θέμα. Αν δεν έχετε την απάντηση, δεν την γνωρίζετε, γραπτά να μου απαντήσετε για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αξιολογήσει. Κάθε πρόγραμμα αξιολογείται ατομικά από ό,τι γνωρίζω. Αλλά στι περιπτώσει συλλογή αποθήκευση άνθρακα, κάποια από αυτά τα προγράμματα, το ξέρω γιατί προέρχονται από τη δική μου περιφέρεια, αφορούν συνδεόμενα σε ένα σύνδεσμο προγραμμάτων ε, τμήματα. Λαμβάνεται υπόψη αυτό το clustering, αυτή η συνένωση ως συνδυασμός ε, όταν αξιολογείται τέτοιου είδους εγχειρήματα για την κοινή, ας το πω έτσι, ε, αποθήκευση και μέσα σε ένα κοινό σύστημα. Σας ευχαριστώ. Chairman, and, uh, και ευχαριστώ πραγματικά γιατί θέσατε τα αριθμητικά μεγέθη σε αναλογία και μια, ένα πλαίσιο. Είναι πολύ επικοδομητικό. Αλλά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι η ένταξη των κλιματολογικών, κλιματικών θεμάτων στον προϋπολογισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε υπέρ της μείωσης ε, των επιδοτήσεων σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα και από ό,τι γνωρίζουμε σε σχέση με τέτοιες, ε, τέτοια χειρήματα η Σλοβενία, Πολωνία που υπάρχουν δεν έχουμε φτάσει στον τελικό στόχο αλλά αυτό είναι το ένα τμήμα. Το άλλο είναι η ένταξη των θεμάτων, των κλιματικών θεμάτων στον προπολογισμό και στις δράσεις. Είμαστε πρόθυμοι να δούμε αυτή τη συνιστόσα, αν είναι επιζήμιες για τις κλιματικές αλλαγές ε, αναφερθήκατε σε σχέση με αυτή τη νέα γενεά. Όταν επικεντρωθούμε στις μεταφορές βλέπουμε 50% των δράσεων της ΕΤΕ πάνε στις οδικές μεταφορές και 10% μόνο στις εναέριες μεταφορές. Αν δείτε ποια ποσά διατίθενται στις δημόσιες μεταφορές σε αστικά κέντρα, τότε είναι ακόμα πολύ μικρότερα, πολύ μικρότερα. Και αν δείτε την αναλογία και την ισορροπία για τα ποσά για τις κεντροανατολικοευρωπαϊκές χώρες, θα δείτε το, τα δύο τρίτα πάνε στις οδικές μεταφορές. Μεγάλη δυσαναλογία. Και ως προς αυτό καλό είναι να επικεντρωνόμαστε στην αποδοτικότητα της ενέργειας και στα ανανεώσιμα όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά δεν έχουμε φτάσει στο να εντάξουμε τα θέματα του κλίματος, που είναι ουσιοδέστατο θέμα, στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον εντάσσονται τα θέματα κλίματος στα εγχειρήματα και στα σχέδια της ε, ΕΤΕ και να ξέρουμε σε σχέση με το 20 ε, ή και λιγότερο ε, του 20% και στις ευρωπαϊκές χώρες είναι ακόμα μικρότερο. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των ευρύτερων αυτών εγχειρημάτων για τις εναέριες μεταφορές και τις οδικές μεταφορές. Πολλά κονδύλια διατίθενται προς αυτήν την κατεύθυνση των οδικών μεταφορών. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λοιπόν. Mm. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βέμπερ παρακαλώ. Ρίχαρτ Βέμπερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η ερώτησή μου στοχεύει σε μια παρόμοια κατεύθυνση. Και μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται στην τράπεζά σας. Είσαστε μια τράπεζα με ειδικού όρους και προϋποθέσεις, με ένα ειδικό κεφάλαιο ευθύνης. Είσαστε όμως μια τράπεζα παρόλα αυτά. Πώς λαμβάνετε ε, υπόψη, πώς διαμορφώνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων, με ποια κριτήρια χρηματοδοτούνται προγράμματα. Δεν θέλω να πω προάγονται, αλλά χρηματοδοτούνται κατά πόσον διαδραματίζει η αηφορία και η εξέταση της αηφορίας ένα ρόλο που αναφέρθηκε από πολλούς συναδέφους ε, ως ε, θέμα και το climate mainstreaming θέλω να αναφέρω αυτή την πτυχή και πολλά άλλα συναφή που εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Ποιο ποσοστό των αποφάσεων ε, αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος όταν πρόκειται συνολικά για θέματα περιβάλλοντος. Πώς εντάσσονται αυτά και κυρίως με ποια κριτήρια λαμβάνονται οι αποφάσεις τι γίνεται ακριβώς σε σχέση με αυτές τις διαδικασίες λήψης απόφασης και πώς μετά αυτά ελέγχονται. Το δεύτερο αφορά τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας της τράπεζάς σας. Άκουσα ότι μεγάλα προγράμματα υποδομών δεν υποβάλλονται πλέον στην ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διότι καλύτερα χρηματοδοτούνται από την ελεύθερη ε, αγορά για παράδειγμα η σύραγγα του Μπρένερ, η καινούρια σύραγγα. Η ελεύθερη αγορά κεφαλαίων είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, είναι καλύτερη για τους όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά τα επιτόκια και τους όρους χρηματοδότησης από την ΕΤΕ. Τι είναι ε, το ενδιαφέρον για σας ε, για να διατίθενται τα κονδύλια. Είναι προγράμματα τα οποία στην ε, ίδια την ελεύθερη αγορά μπορούν να διασφαλίσουν κονδύλια και τι θα κάνατε εσείς και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, για να υπάρξει δυνατότητα δυναμικού διανομής ε, στην ε, Ευρώπη. Τα δίκτυα υποδομής στον τομέα των ενεργειακών θα πρέπει να επεκταθούν σε ιδιαίτερο βαθμό θέτετε εσείς κέντρο βάρους σε αυτό ή δεν βρίσκονται, δεν εξαρτώνται αυτοί οι οποίοι θα ασχοληθούν με το δίκτυο διανομής από την ΕΤΕ. Και τέλος παρακαλώ ο Κονή le président Ευχαριστώ. Απευθύνομαι σε εσά και σε σχέση με το ε, θέμα της ε, ομάδας ε, για τα θέματα των αστικών κέντρων και ως πρώην μέλος της ε, η Επιτροπής Περιφερικής Ανάπτυξης στην Ευρω... στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενδιαφέρομαι άμεσα και ιδιαίτερα και είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη για τα θέματα ε, αυτά στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στην έκθεση του 2010, δηλαδή πέρυσι, φαίνεται ότι 15 κεφάλαια Τζέσικα αφορούν 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για την αηφόρο ανάπτυξη αστικών κέντρων ε, πόλεων κτλ. Το ερώτημα είναι το Τζέσικα θα συνεχιστεί ως εγχείρημα για την προαγωγή ε, προγραμμάτων και σχεδίων για την μείωση των εκπομπών ρήπων ε, θερμοκηπίου. Πιστεύετε ότι αυτή η υποστήριξη για την αηφορία στην ανάπτυξη με δάνεια και πιστώσεις ε, για την επίτευξη της μείωσης των εκπομπών ρήπων και με γενική υποστήριξη θα μπορούσε να συνεχιστεί για όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αναφέρατε πιο πριν ότι στον οδικό χάρτη 2050 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι ετήσια θα απαιτούν ε, πολλά δισεκατομμύρια ευρώ και από πλευράς ε, του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μεγεθύνεται και κάποιες κυβερνήσεις ανθίστανται, με τα ευρωομόλογα θα μπορούσε κανείς να προχωρήσει με ένα τρόπο διασφάλισης κονδυλίων εκτός προϋπολογισμού. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό από πλευράς της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με τα ευρωομόλογα, project bonds, ε, ομόλογα έργου τα αποκάλεσαν αυτά. Ε, πώς θα μπορούσε αυτό για την χρηματοδότηση του περιβάλλοντος να δράσει. Έχουμε αρκετά κονδύλια ή χρειάζονται καινούρια. Ευχαριστώ. Αυτά είναι κάποιες από τις ερωτήσεις ε, που αναφύονται σε σχέση με αυτά τα θέματα. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που τίθενται και πρέπει να απαντηθούν. Διαφορετικά και σε ερωτήσεις. Να ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση που ε, εσείς διατυπώσατε για να αποφύγουμε παρανοήσεις. Πολλά έχουν αναφερθεί για τα ευρωομόλογα. Πρέπει να γίνει ένας σαφής διαχωρισμός, σαφής διαφοροποίηση μεταξύ διαφορετικών τύπων ευρωομολόγων. Τρεις διαφορετικοί τύποι υπάρχουν. Πρώτα τα, τα ε, ομόλογα δολαρίου, αυτά τα οποία όταν γινόταν λόγο σε σχέση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα για την ενέργεια και τη μεταφορά από τον Ζακ Ντελόρ είχαν ε, αναφερθεί. Χρηματοδότηση ομολόγων της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη, ας το πω έτσι, προσέγγιση ομολόγων που διασφαλίζονται και κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν κάτι το οποίο αρνήθηκε το Συμβούλιο, όπως θα γνωρίζετε. Η δεύτερη προσέγγιση ευρωομολόγων, τα ομόλογα Juncker όπως αποκαλούνται, διότι στόχευαν μεταξύ άλλων από τον Λουξεμβούργιο Πρωθυπουργό ε, Jean-Claude Juncker θα ε, χρηματοδότησε από τα διαφορετικά κράτη-μέλη με διάφορους τύπους που είχαν προταθεί. Αλλά ουσιαστικά θα ήταν ομόλογα που τα κράτη-μέλη θα εξέδιδαν με υπηρεσίες που θα τα εξέδιδαν για το λογαριασμό αυτών των κρατών μελών. Τώρα, το, ο τρίτος τύπος, ας το πω έτσι, είναι αυτά τα οποία μπορούμε να τα αποκαλέσουμε ομόλογα Μπαρόζο, γιατί προτάθηκαν από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένα τελείως διαφορετικό είδος ομολόγων δεν θα, τα εξέδιδαν τα κράτη-μέλη ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από οι διαχειριστές, οι ιδιώτες διαχειριστές ε, σχεδίων και προγραμμάτων. Έκδοση ομολόγων για την διασφάλιση κονδυλίων για μεγάλα προγράμματα υποδομής. Τι γίνεται εδώ, ποιο είναι ο λόγο. Ο λόγο είναι ότι δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε όλο το εύρο των έργων υποδομών με δημόσια χρηματοδότηση. Θα ήταν λοιπόν οι θεσμικοί επενδυτέ εκείνοι που θα συμφωνούσαν να δανειοδοτήσουν με κονδύλια μακροπρόθεσμα τέτοιου είδου έργα υποδομών. Και για την διασφάλιση τους, για αυτοί οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές, α το αποκαλέσουμε έτσι, θα έπρεπε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για την αξιολόγησή τους σε συγκεκριμένες κλίμακες ή βαθμίδες πιστοληπτικής αξιοπιστίας. Και έτσι θα έπρεπε να δούμε ότι οι αρχές θα είχαν ένα μικρότερο τμήμα κεφαλαίου που θα διατίθετο και οι ιδιωτικοί επενδυτές θα είχαν ένα πολύ μεγαλύτερο ε, μέρος ή τμήμα. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά αυτές είναι οι τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις για τα ευρωομόλογα. Και η πιο πρόσφατη προσέγγιση είναι αυτή όπου οι ιδιώτες επενδυτές, οι ιδιωτικοί επενδυτές ε, θα ήταν οι πιο ευπρόσδεκτοι και θα εμπλεκόντουσαν περισσότερο. Σε σχέση με τα εμπόδια που ρωτήσατε, που ίσως υφίστανται σε σχέση με την ΕΤΕ, ουσιαστικά θα έλεγα, ο κύριος ρόλος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες και οι κανονισμοί για τα χρηματοοικονομικά θέματα και για ε, τις λειτουργίες τις χρηματοοικονομικές θα έπρεπε να μπορούν να διασφαλίσουν αυτού του είδους τις κοινέ δράσεις και να τις διευκολύνουν κιόλας. Δεν θέλω να επισέλθω σε τεχνικής, φύσης ε, ε, τεχνικού χαρακτήρα λεπτομέρειες, αλλά σε σχέση με το ετήσιο χρηματοοικονομικό πλαίσιο, με την έγκρισή του θα ζητηθεί από το Ευρωκοινοβούλιο να συζητήσει αυτούς τους χρηματοοικονομικούς κανονισμούς και διατάξεις. Μέσα από μια τέτοια εταιρική σχέση στρατηγικής, ένα τέτοιο πολιετές στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να διευκολύνει τις διαδικασίες. Να επισέθω στι πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αναφέρατε το Ελένα. Είναι ένα πρόγραμμα τεχνικής αρρωγής που θα βοηθά την κατάρτιση και συγκρότηση προγραμμάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Είναι πιλωτικό αυτό το πρόγραμμα, αλλά τα πρώτα αποτελέσματα είναι αρκετά θετικά. Στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε ποιο earmarking, ποιο προκαθορισμός κονδυλίων μέσα στον προϋπολογισμό θα πρέπει να επιτυγχάνεται. Για το 300, AER 300, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω για την αξιολόγηση, την μέθοδο αξιολόγησης. <clears throat> μπορώ να επιβεβαιώσω σε σχέση με αυτήν ότι λάβαμε 78 αιτήματα από κράτη-μέλη και καθώς γνωρίζετε η ΕΤΕ έχει μία περίοδο ενέάμινη εννέα μηνών για την ε, υποβολή των συστάσεών της ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μηνή αυτή περίοδος δεν είναι ιδιαίτερα ευρεία, δεν είναι πολύ μεγάλη για αυτό το έργο. Κάνουμε βέβαια προσπάθεια να τηρήσουμε αυτά τα χρονοδιαγράμματα, αυτά τα χρονικά πλαίσια. Αναλύοντας αυτά τα προγράμματα και τα σχέδια, λαμβάνουμε υπόψη και αξιολογούμε και το clustering effect, όπως ανέφερε η κυρία Μακάβεν πιο πριν δηλαδή τις επιπτώσεις ε, κοινών προγραμμάτων ή από κοινού ομάδων. Και έχει απόλυτο δίκιο σε σχέση με την παρέμβαση ε, ο συνάδελφος πιο πριν αληθεύει ότι πρέπει να έχουμε κάποιο βαθμό ελαστικότητας για να είμαστε αποτελεσματικοί. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Επακούμε σε αυτό. Διότι αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα ζητήματα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ευαίσθητα θέματα για την αγορά. Όμως θα ήταν προς το συμφέρον όλων να έχουμε αρκετό πλαίσιο για ελαστικότητα ώστε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μπορεί να διασφαλίσει ότι θα είναι αποτελεσματικά τα θέματα τα οποία θα α, ρυθμίσει με αυτόν τον τρόπο. Euh, δεν θα πρέπει να παίρνει κανείς τις μετρητής αυτά τα οποία λένε. Ρόλος τους είναι να ασκούν κριτική στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων, χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά. Γι' αυτό αυτό δεν σημαίνει ότι βασίζονται κάπου, αν και δεν θα πρέπει να αγνοηθεί η κριτική που ασκούν. Για το τμήμα της παραγωγής ηλεκτρισμού που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα υπήρξε μια πολύ σημαντική αλλαγή θα έλεγα Ήδη από το 2000 το τμήμα, το 2000 το τμήμα των ορεικτών καυσίμων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά το 2007 εμείς προχωρήσαμε σε αλλαγές, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν έχουμε δική μας πολιτική, υποστηρίζουμε την πολιτική που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν πράγματι η καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών έγινε μια πραγματικότητα, έγινε και για μας και γι' αυτό από το 2007 υιοθετήσαμε σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου μια πολιτική θα έλεγα αλλαγή και υπήρξαν πολύ πιο αυστηρά κριτήρια για χρηματοδότηση εγκαταστάσεων με ορυκτά κάψιμα και γι' αυτό το τμήμα αυτό έχει μειωθεί ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κατηγορούμε την τράπεζά μου για το τι γινόταν στο παρελθόν ενώ έχουμε αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Θα επανέλθω σε υπόλοιπα, σε άλλα θέματα αργότερα. Θέσατε επίσης ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Έχετε απόλυτο δίκιο όταν υποστηρίζετε ότι δεν μπορούμε να περιοριστούμε λέγοντας ότι χρηματοδοτούμε ανανεώσιμες πηγές και δεν κάνουμε τίποτα άλλο για ό,τι άλλο. Είναι αλήθεια ότι όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτεί η τράπεζά μου πρέπει να εξεταστούν και σε επίπεδο περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σε επίπεδο κυρίως εκπομπής καυσαερίων θερμοκηπίου. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε εμείς να δούμε ποιο είναι το ίχνος σε άνθρακα όλων των χρηματοδοτήσεων στην οποία έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αν θέλει η Επιτροπή σας, κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να είχαμε μια συζήτηση σε βάθος. Τίθενται ορισμένες μεθοδολογικές δυσκολίες εδώ. Συνεργαζόμαστε σε συνεργασία και με άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως την Παγκόσμια Τράπεζα, και ανταλλάσσουμε τις εμπειρίες μας στον τομέα αυτό. Κάναμε όμως κάποιες προσπάθειες σε όλα τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν το 2009. Και από ό,τι φαίνεται κάναμε ένα έλεγχο λοιπόν και από ό,τι φαίνεται, είμαι λίγο επιφυλακτικός εδώ, ότι τελικά ο απολογισμός είναι θετικός. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μία μείωση κατά 2, ε, κατά 2 εκατομμύρια 400 τόνους ε, διοξιδίου του άνθρακα κατέτος. Ο αριθμός ε, σε επίπεδο ακρίβειας ίσως να μην είναι σωστός αλλά εμείς είμαστε υπέρ αυτού του mainstreaming, δηλαδή εξετάζοντας όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουμε μία ανάλυση των συνεπειών σε επίπεδο εκπομπών, αναπτύσσουμε μία μεθοδολογία η οποία νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα προχωρημένη σχετικά με το περιεχόμενό της και επ' αυτών των βάσεων για το 2009 όπου έχουμε κάνει σε σύνολο εξέταση της κατάστασης το αποτέλεσμα είναι ελαφρά θετικό. Αλλά η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί. Θέσατε ερωτήσεις και για τις μεταφορές επίσης. Δεν έχουμε χρόνο να μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά αν δει κανένα τα τελευταία στοιχεία θα δει ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης των σιδηροδρόμων και κυρίως των αστικών συγκοινωνιών μετρό κτλ. Βέβαια θα πρέπει να λάβουμε και άλλες εξελίξεις υπόψη ε, λόγω της προσπάθειας που κάνουμε να ακολουθήσουμε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσατε για την αεροναυτική. Εμείς δεν χρηματοδοτούμε πλήρως τέτοιου είδους εταιρείε ούτε και αεροδρόμια παρακάτω από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αεροδρόμια σε υπερηφέρειες απόμακρες ή αν οι επενδύσεις επιτρέπουν να μειωθεί η εκπομπή καυσαερίων στην περιοχή. Είναι μια στάση που έχουμε την οποία αμφισβητούν πάρα πολλές χώρες και ασκούν κριτική στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το ότι χρηματοδοτεί τον αεροναυτικό τομέα πολύ πιο περιοριστικά από ό,τι στο παρελθόν. Κύριε Σέμπερ, θέσατε ερωτήσεις και για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην τράπεζά μας. Ε, σχηματικά θα το πω, γίνεται μια πρώτη ε, επιλογή σε επίπεδο ακριβώς επιλεξιμότητας να δούμε αν δηλαδή συνεισφέρει η πρόταση στην επίτευξη στόχων της πολιτικής ένωσης. Αν είναι επιλέξιμο ένα πρόγραμμα, τότε το εξετάζουμε τεχνικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά και φυσικά χρηματοδοτικά. Είμαστε λίγο περίεργη τράπεζα γιατί έχουμε πάνω από 150 μηχανικούς που εξετάζουν τα τεχνικά κομμάτια των προγραμμάτων και κυρίως τον σεβασμό των περιβαλλοντικών κανόνων. Στη συνέχεια το πρόγραμμα υποβάλλεται στον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κάνει μια διυπηρεσιακή θα έλεγα εξέταση και φυσικά η υπηρεσία που ασχολείται με το περιβάλλον, που ασχολείται με το περιβάλλον είναι βασικός πρωταγωνιστής αυτής, της, αυτού του σταδίου και στη συνέχεια εφόσον είναι θετική άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο το πρόγραμμα. Αυτά περιληπτικά. Τώρα, ε, ποιο είναι το ενδιαφέρον προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ κάποιοι άλλοι βρίσκουν καλύτερους όρους ε, στην αγορά. Γιατί όχι, αυτή είναι η αρχή της επικουρικότητας, αλλά αυτό μου φαίνεται μάλλον εξαίρεση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τρέφεται κανένα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και λόγω των τεχνικών αναλύσεων τις οποίες προανέφερα, γιατί περιμένει ο ιδιωτικός τομέας να πάρουμε αποφάσεις, είναι σαν μια ετικέτα ποιότητας το αν το χρηματοδοτούμε ή συγχρηματοδοτούμε. Ακολουθούν οι εμπορικές τράπεζες και ο δεύτερος λόγος για τον οποίο προσφεύγουμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι η διάρκεια των δανειοδοτήσεών μας. Εμείς δανειοδοτούμε για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από τις εμπορικές τράπεζες, 25 χρόνια ή 30 χρόνια, πολλές φορές και περισσότερα. Και ο τρίτος λόγος πάρα πολύ συχνά είναι ότι μπορούμε να προσφέρουμε σε επίπεδο επιτοκίων καλύτερους όρους, γιατί εμείς δανείζουμε από τις, δανειζόμεθα από τις χρηματαγορές ε, με καλούς όρους γιατί έχουμε 3α, μετά έχουμε το, το ενδιάμεσο κόστος για να καλύψουμε τη λειτουργία μας σαν ένα κίνδυνο κάλυψης κινδύνου, και φτάνει κανείς στο να προτείνει, θα έλεγα, ύψη ε, επιτοκίων ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Ε, η κυρία Χάουκεν για το Τζέσικα ειλικρινά ε, αυτή η χρονιά θα είναι καθοριστική για τον Τζέσικα αγαπητή κυρία θα πρέπει να αποδείξουμε ότι το Τζέσικα λειτουργεί σωστά χρειάστηκε πολύς χρόνος γιατί ήταν ένα καινούριο πρόγραμμα και έπρεπε να ρυθμιστεί η λειτουργία του ε, το Jessica είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ένα τμήμα των διαφορετικών ταμείων για να δημιουργήσουν ε, εταιρείε χρηματοδότησης προγραμμάτων ε, ανανέωσης και ανακαίνησης περιοχών στο εσωτερικό των πόλεων. Ε, είπατε ότι υπάρχουν 15 τέτοια ταμεία τα οποία βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας, κάποια λειτουργούν ήδη, αλλά στο τέλος του χρόνου θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και θα πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό της προσπάθειας του χρόνου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Μαστάτη, είχε πολύ ενδιαφέρον η παρουσίασή σας. Αναφερθήκατε στα θέματα με πολύ μεγάλη. Ξέχασα μια ερώτηση, λέει ο κύριος ε, Δεν θα πρέπει να αφήσουμε κενά, λέει ο Πρόεδρος. Είναι κάτι το οποίο δεν σχετίζεται άμεσα με αυτό που συζητάμε σήμερα. Με ε, λίγα λόγια θα πω εδώ. Είμαι στην διάθεση της Επιτροπής σας αν θέλετε μεγαλύτερη συζήτηση. Πρόκειται για ένα σχέδιο αυτό το οποίο θέσατε, το οποίο χρηματοδοτήσατε και το οποίο έχει σαν στόχο την μείωση της, εκπομπής ε, ε, καυσαερίων Déjà diminué de plus Τα καυσαέρια που προέρχονται από θείο. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε, είναι ένα πρόβλημα φοροδιαφυγής. Φαίνεται ότι δημιουργήθηκαν κάποιοι μηχανισμοί που οδηγούν τελικά στη μετακίνηση του κέρδους εκτός της χώρας και στην φοροδιαφυγή ε, τουλάχιστον σε επίπεδο εθνικής φορολογίας. Όταν το μάθαμε ε, προειδοποιήσαμε την ΟΛΑΦ που καταπολεμά την απάτη και, ε, και ξεκινήσαμε και τη δική μας έρευνα. Πήγαμε και επί τόπου, η μονάδα μας ενώ η ερευνητική. Στην αρχή δεν είχαμε και πολύ ε, πολύ ιδιαίτερη καλή συνεργασία από την εταιρεία. Αναγκαστήκαμε να την απειλήσουμε ότι θα ζητήσουμε επιστροφή του δανείου ε, εκ των προτέρων. Από τότε τα πράγματα πάνε καλύτερα, η έρευνα εξελίσσεται συνεχώς. Αλλά εάν η κατηγορία επιβεβαιωθεί, τότε σε αυτή την περίπτωση θα ζητήσουμε την πλήρη επιστροφή των ποσών έδωσα οδηγίες στις υπηρεσίες μου και για άλλους λόγους να μην δέχονται αιτήσει χρηματοδότησης που προέρχονται από την εταιρεία Glencore ή από μία θηγατρική. Αυτό είναι θέμα διακυβέρνησης εταιρικής που ξεπερνά την επένδυση στο Μοπανί. Είναι θέμα, διαβάστε τη Financial Times την προηγούμενη εβδομάδα, θα δείτε τα προβλήματα με την Glencore, ε, και γι' αυτό ακριβώς δεν δεχόμαστε ε, θηγατρικές εταιρείες ή τη συγκεκριμένη εταιρεία να ζητά χρηματοδοτήσεις από μας. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας τα επόμενα χρόνια. Το Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί από κοντά τις δραστηριότητές σας με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα σας στηρίξουμε εφόσον ακολουθείτε την σωστή γραμμή. Καλή επιτυχία λοιπόν και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ και την επιμελητία. Στις... Αύριο το πρωί